Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω να καθίσετε. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχουμε τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο σήμερα μαζί μας για το απόγευμα, αλλά στις 4 και 35 το αργότερο πρέπει να αποχωρήσει. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να προλάβουμε μέσα στο χρόνο που έχει να μας διαθέσει. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε προβλέψει για σήμερα είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο για την εφαρμογή των τριχών των μέτρων και τις νέες προτάσεις Κομισιόν από τις 7 Ιουνίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω κατευθείαν το λόγο στον Επίτροπο να μας κάνει μια παρουσίαση και μετά θα δώσω το λόγο στους συντονιστές να κάνουν ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά θα τους απαντήσει ο Επίτροπος και μετά θα κάνουμε ένα καινούριο γύρο ερωτήσεων για τα άλλα μέλη και μετά θα ξεκινήσει και η συζήτηση. Κύριε Αβραμόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη χαρά για μας που ξαναέρχομαι εδώ και πάλι. Έχουν περάσει τεσσερά μήνες από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε για τελευταία φορά στα πλαίσια του διαλόγου που κάνουμε τον Ιανουάριο και μας δίνει μια ευκαιρία πρώτα απ' όλα να συζητήσουμε τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, την πρόοδο που έχουμε πετύχει σε κάποιους φακέλους κλειδιά και βέβαια το τι ακόμα μένει να πετύχουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω Πρώτα απ' όλα αναφερόμενος στο θέμα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και θα σας κάνω μια πολύ γρήγορη ενημέρωση για την πρόοδο που έχουμε για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το θέμα αυτό συζητήθηκε την Παρασκευή από τους Υπουργού Εσωτερικών και σήμερα η Κομισιόν εξέδωσε μια δεύτερη έκθεση για το πώς τρέχει η εφαρμογή της συνθήκης αυτής. Η συμφωνία λοιπόν της ε, Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε πολύ έντονα τις μεταναστευτικές ροές. Οι αφήξεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί ριζικά, αλλά ακόμα είναι μια πρόκληση για το δυναμικό υποδοχής που έχει η χώρα. Ο ρυθμός της μετεγκατάστασης έχει διπλασιαστεί σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Έχουμε δηλαδή 700 περίπου Έχουμε επίσης δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους που περιμένουν ακόμα την ευκαιρία στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Για να μοιραστούν περισσότερο αυτή την ευθύνη μεταξύ τους τα κράτη-μέλη, θα πρέπει με το θέμα αυτό να ε, εργαστούν πιο γρήγορα και να πάρουν κόσμο και από την Ιταλία και από την Ελλάδα και να βοηθήσουν τις δύο αυτές χώρες. Οι προσπάθειες που γίνονται για να μεταφερθεί κόσμος από την Τουρκία στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης έχουν ε, ε, πετύχει αρκετά. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, και με, το, με την εξέταση των αιτήσεων ασύλου ε, στην Λέσβο. Έχουμε και την εξέταση ε, αιτήσεων ασύλου που θα πρέπει να ξεκινήσει στα άλλα νησιά, γιατί στη Λέσβο στο έχει ξεκινήσει, όπως επίσης και για κατηγορίες πέραν αυτή των σύρων. Η η Ελλάδα έχει στηριχθεί και νομίζω πως θα πρέπει να συνεργαστούμε και εμείς πολύ σαν αναμετρήτες χώρες, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία με τους εταίρους μας για να έχουμε καλύτερη συνεργασία και για την επανεισδοχή και για τις επιστροφές. Θα πρέπει να πάψουμε να ε, προσποιούμεθα πως οι σχέσεις μας ε, ακολουθούν το μοντέλο business as usual. Δηλαδή, ε, μια φυσιολογική ροή της κατάστασης όταν κάποιοι από εμά ε, και κάποιοι από τους εταίρους μας δεν σέβονται την υποχρέωσή τους να ε, δεχθούν πίσω τους υπηκόους τους. Την τελευταία φορά που τα είπαμε στην Ολομέλεια μιλήσαμε για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και ελπίζουμε πως το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη νέα προσέγγιση θα την στηρίξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτή τη νέα έννοια. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συντονισμένες προσπάθειες που κάνουμε, να πατάξουμε τα δίκτυα των ε, πασαδόρων που αυτή τη στιγμή στοχεύουν στο πιο ευάλωτο κομμάτι αυτού του πληθυσμού και να δούμε και τι γίνεται και με την κατάσταση των ε, μεταναστών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ στο Κοινοβούλιο για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που κάνετε σε αυτό το θέμα. Και να σας πω πως υπάρχει το πρόβλημα των λαθρέων εισόδων. Έχουμε και το πρόσφατο ψήφισμα για την εφαρμογή ε, της ε, οδηγίας κατά του τράφικιν, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου. Επίσης, ε, περιμένω και την εγκρίση του ψηφίσματος για τη μάχη για την πάταξη του τράφικινγκ ε, με ανθρώπους ε, στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της σφαιρικής προσέγγισης που ακολουθούμε που είναι η μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 4 Μαΐου παρουσιάσαμε το πρώτο σχέδιο και νομίζω ότι έφτασε πια η ώρα για ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα που θα βασίζεται σε κοινού κανόνες και σε μια δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Με τις προτινόμενες αλλαγέ που θα εισάγουμε στο σύστημα θα ενισχύσουμε τη Eurodac και η ΕΑΣΟ θα γίνει μια πραγματική ε, ευρωπαϊκή υπηρεσία για το άσυλο. Με τον τρόπο αυτό θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς αυτή τη στιγμή στείλουμε τις δομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργούμε τα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι απαραίτητα για ένα συνολικό σφαιρικό σύστημα. Εγώ βασίζομαι εδώ στον κύριο Κύρκοφ, στον κύριο Μίντερμιλ και στην κυρία Βίξτρομ που είναι οι, οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές για τα θέματα αυτά ε, βασίζομαι σε εσά για να με στηρίξετε έτσι ώστε να έχουμε μια ομαλή πορεία έγκρισης για αυτό το φάκελο. Το δεύτερο πακέτο που είναι εξίσου φιλόδοξο ε, θα περάσει τον Ιούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις επίσης για να έχουμε ε, καλύτερη ενσωμάτωση μεταναστών από τρίτες χώρες με καλύτερη οικονομική και κοινωνική συνεισφορά από τα άτομα αυτά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για μια πολύ καρποφόρο συζήτηση που κάναμε την περασμένη Τρίτη για το νέο σχέδιο δράσης που μόλις εγκρίθηκε για την ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών, όπως επίσης και για το προτινόμενο όραμα που παρουσιάσαμε για τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία. Ε, εμείς θα στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ε, και τις επιχειρήσεις τη στιγμή που θέλουμε να προσελκύσουμε υψηλά κατευθυσμένα στελέχη από τρίτες χώρες για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στην οικονομία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Οι δύο αυτέ πρωτοβουλίες αποτελούν κομμάτι της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για την νόμιμη μετανάστευση. Νομίζω ότι αυτό το είπα ξεκάθαρα την περασμένη εβδομάδα. Είναι ακριβώς προς το συμφέρον όλων μας να δείξουμε την πολιτική βούληση έτσι ώστε το θέμα αυτό να τεθεί ως προτεραιότητα. Να έχουμε νόμιμη μετανάστευση, να έχουμε ενσωμάτωση των μεταναστών και παράλληλα να έχουμε και δράσεις οι οποίες αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες των ε, προσφύγων. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο δυνατή και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε ένα από τα θέματα τα οποία εγώ θεωρώ ζωτική σημασία και ξέρω πως οι περισσότεροι από εσάς θα συμφωνήσετε μαζί μου ε, που είναι οι προσπάθειες για να διατηρήσουμε την ακαιρεότητα του χώρου Σέγγεν. Ελπίζω πως θα συμφωνήσουμε για το θέμα αυτό μέχρι τα τέλη ε, του μήνα για την ακτοφυλακή και τη συνοροφυλακή της Ευρώπης. Η νέα αυτή η υπηρεσία θα στηρίξει τα ευρωπαϊκά σύνορα, θα τα εξασφαλίσει, θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τα θέματα ε, τα μεταναστευτικά και θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ασφαλή. Ένα τελευταίο θέμα που είναι επίση εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως αυτές οι δύο νέες υπηρεσίε θα εξασφαλίσουν την αρχή της ελεύθερης μετακίνησης μέσα στο χώρο Σέγγεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εισηγητές και στα μέλη όλων των ομάδων για τις πάρα πολύ εντατικές προσπάθειες που έκαναν για ένα θέμα δύσκολο με ασφικτικό χρονοδιάγραμμα. Τώρα, ας έρθω στις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του μηχανισμού απαλλαγής από τις θεωρήσεις και ε, την απελευθέρωση για την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Κωσυφοπαίδιο και την Τουρκία. Για την πρώτη πρόταση η συζήτηση Πρέπει να σας πω ότι προχωράει γρήγορα. Χαιρετίζω την προτεραιότητα που έχει δώσει το φάκελο αυτό το Κοινοβούλιο και είμαι πεπισμένος πως αυτός ο μηχανισμός θα συμφωνηθεί, ο μηχανισμός αναστολής από τους συνομοθέτες χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά για τον μηχανισμό αυτό ε, θα πρέπει να πω το εξή. Δεν θα πρέπει το ότι το συζητάμε να παρακολύσει τη συζήτηση για την απελευθέρωση, για τι θεωρήσει για Γεωργία, Ουκρανία, ε, και Τουρκία. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που την Παρασκευή το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει για τη Γεωργία. Κάθε χώρα θα πρέπει να εξεταστεί μεμονωμένα και να αποφασιστεί βάσει στα δικά τη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Χαίρομαι που υπάρχει πολιτική δέσμευση από το Συμβούλιο για το φάκελο αυτό και βέβαια θα ήθελα να ε, στηριχθώ σε εσά για να πετύχουμε απτά αποτελέσματα και ε, ε, επιτυχίες. Τώρα, για την αμοιβαιότητα για τις θεωρήσεις με τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ, έλαβα και κατέγραψα την επιστολή ε, που έλαβα από τον από τον πρόεδρο και πρέπει να σας πω πως ε, γνωρίζουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και όπως είδατε στις ανακοινώσεις μας του Απριλίου, ξέρουμε ότι υπάρχουν αρνητικές πολιτικές και οικονομικές ε, ε, συνέπειες από οποιαδήποτε αναστολή. Η αμοιβαιότητα στις θεωρήσεις συζητήθηκε σε μια υπουργική ε, συνάντηση, μια συνάντηση υπουργικού επίπεδου με τη ΣΥΠΑ στις 2 Ιουνίου και πρόσφατα συνάντησα τον Ζαν Μακάλαν που είναι ο Καναδός Υπουργό για τη Μετανάστευση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχω σκοπό να εντατικοποιήσω τις επαφές αυτές σε όλα τα επίπεδα. Εμείς συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε πλήρη αμοιβαιότητα για όλα τα κράτη-μέλη για τις θεωρήσεις και με τη ΣΥΠΑ και με τον Καναδά. Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει όλοι μαζί για τα θέματα ασφάλειας αναγνωρίζεται από τους εταίρους μας ε, απερίφραστα και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και τις ζητήσεις που κάνουμε. Το πλαίσιο το οποίο παρουσιάσαμε για μια πραγματική και αποτελεσματική ένωση ασφάλειας στην Ευρώπη είναι η κατεύθυνση ακριβώς προς την οποία πρέπει να κινηθούμε για να πετύχουμε αυτό που σας περιγράφω. Γιατί η εσωτερική ασφάλεια ενός κράτους μέλους είναι ακριβώς και η εσωτερική ασφάλεια ολόκληρης της Ένωσης. Έχουμε σαφείς προτεραιότητες για το μέλλον και αυτές είναι, καταρχήν, να βελτιώσουμε το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Η διασύνδεση και η διασυνδεσιμότητα μεταξύ βάσεων με δεδομένα ασφαλείας. Και όλοι οι αξιωματικοί ασφάλειας να έχουν τα ίδια τα ανακλαστικά και να μοιράζονται τις πληροφορίες με τους συναδέλφους τους ε, στα σύνορά τους, όπως ακριβώς το κάνουν μέσα στην ίδια την επικράτεια της χώρας τους. Στα πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος ασφάλειας, ελπίζω πως... Ε, το κέντρο ε, της ε, αντιτρομοκρατικής στην Ευρώπη και η Europol θα αποτελέσουν τον πυρήνα, τον κόμβο όλων αυτών των προσπαθειών για την αξιολόγηση κινδύνων, για λειτουργικό συντονισμό, όπως επίσης και για ανταλλαγή πληροφοριών. Τους δώσαμε επιπλέον πόρους για το 2016. Και με τη δική σας στήριξη και με τη δική σας ενισφορά καταφέραμε να δώσουμε στη Europol ένα νέο νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της και στην αποστολή της. Έχουμε και την οδηγία για τα δεδομένα των επιβατών, την PNR, και θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και γρήγορα. Δεν ε, θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω στα κράτη-μέλη. Εμείς στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα κράτη-μέλη. Οι εμπειρογνώμονέ μα ε, συναντιόνται μαζί του για να συζητήσουν ποιε είναι οι προκλήσει. Τώρα για τα πυροβόλα όπλα. Εκεί έχουμε τη γενική προσέγγιση στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο την, ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι μόλι η αντίστοιχη εδώ Επιτροπή ε, τελειώσει με τα δικά τη θέματα. Και έχει να κάνει το θέμα αυτό και με την ασφάλεια αλλά και με την εσωτερική αγορά. Η σφαγή στο Ορλάντο νομίζω απέδειξε επώδυνα για μία φορά ακόμα πως αυτό είναι ε, σοβαρό. Τα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς ε, διασκέδασης ή ε, κυνηγιού θα πρέπει τα καλά σνικόφ, για παράδειγμα, να απαγορευτεί να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μην μπορείς να τα πουλήσεις σε απλούς πολίτες, γιατί χρησιμοποιούνται μόνο για σφαγές, όπως επίσης το R50 που χρησιμοποιήθηκε στο Ορλάντο. Θέλω εσείς να απαγορεύσετε αυτά τα πυροβόλα όπλα στο τελικό κείμενο της νέας οδηγίας. Και σίγουρα μπορώ να βασιστώ σε εσά και κυρίως στην κυρία Χόλμαγερ για να εξασφαλίσουμε πως η μέλους οδηγία για την αντιτρομοκρατία ε, θα βοηθήσει πραγματικά στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Πιστεύω ότι η επόμενη, την επόμενη εβδομάδα η ΛΥΜΠΕ θα εγκρίνει την ε, ε, διαπραγματευτική εντολή και θα ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι. Και εδώ θα πρέπει να φανούμε φιλόδοξοι, κυρίως για την μετακίνηση των τρομοκρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως επίσης οι προσπάθειες που κάνουν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά οπωσδήποτε θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στους νέους κανόνες. Τώρα, για το θέμα ε, της πολιτικής μας κατά των ναρκωτικών, να σας πω πως αυτή τη στιγμή συζητάτε τη νέα προσέγγιση και το νέο ε, ε, ε, πλαίσιο για τις ψυχοτρόπους ουσίες, έτσι όπως τα έχει προετοιμάσει η Ολλανδική Προεδρία. Εμείς θα συνεργαστούμε μαζί σας και με το Συμβούλιο για να το συμφωνήσουμε το θέμα αυτό σύντομα. Τώρα θα ήθελα να στραφώ προς τους τελευταίους πέντε μήνες, να ταινίσω το τι κάναμε τότε και να σας πω πως πραγματικά προδέξαμε πάρα πολύ στα θέματα και της μετανάστευσης και της ασφάλειας, παρόλο που είναι ακόμα πιο πιεστικές οι προκλήσεις, πιο πιεστικές από ό,τι ποτέ. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα στεναρό πλαίσιο για το άσυλο και να ενισχύσουμε τους, ε, τα σύνορά μας Δίνοντα όμως και ελεύθερη πρόσβαση μέσω της απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση σε τους κάποιους ε, πολίτες τρίτων χωρών. Θέλουμε Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να ασκήσουν τα δικαιώματα και τι ελευθερίε τους. Να βρούμε δηλαδή μια σωστή υπηρεσία και πρέπει να σας πω πως οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά και στην Ολομέλεια αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών στο ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απόκριση σε όλες τις προκλήσεις. Αυτή είναι η άουσα και ο δρόμος ε, που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστούμε, Επιτροπέ. Ευχαριστούμε για αυτή σας την εισήγηση. Όπως είπα από την αρχή, θα ξεκινήσω με τους εκπροσώπους των Επιτροπών. Θα ζητήσω από τον κύριο Έγκελ αντί για την κυρία Χολμάγερ. Και μετά θα παριθμίσω τα ονόματα που έχω μπροστά μου στον καταλόγο αγορητών, όσους έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Γιγιόμ, η κυρία Ρεβονταλόν, κυρία Φαγιόν, η κυρία Κινίτσι, η κυρία Γκόμε, ο κύριο Νίντερ Μίλλερ, ο κύριο Πόστο, ο κύριο Βάιντεν Χόσερ, η κυρία Σάινα και η κυρία αυτά από την πλευρά των προσώπων τη της Επιτροπής, θα σας παρακαλέσω να παραμένετε στα δύο λεπτά για να έχουμε και απαντήσεις. Να έχουμε χρόνο δηλαδή για να ακούσουμε τις απαντήσεις. Ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που είπατε ότι είμαστε επίτροποι. Φαντάζομαι ότι εννοείται συντονιστές. Θα ήθελα και εγώ να, να έχω τον τίτλο του επιτρόπου αλλά σε κάθε περίπτωση απέναντι σε ένα πραγματικό επίτροπο πρέπει να εκφράσω την εγγνωμοσύνη μου προς τον Δημήτρη και τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Τέλο πάντων, και να συνεχίσω στα γαλλικά για να έχουμε και την απαραίτητη γλωσσική ποικιλία. Είχα ήδη την ευκαιρία σε αυτή την Επιτροπή όχι απλώς να διαφωνήσω μαζί σας στην Ολομέλεια, αλλά να εκφράσω τουλάχιστον κάποιες ανησυχίες δικές μου σε σχέση με, τη δική μας, με την αναθεώρηση της λογικής μας περί Θα ήθελα να διατηρηθεί η αρχή της απαραίτητης αλληλεγγύης. Όμως γνωρίζουμε ότι την πρώτη φορά αποτύχαμε εκτρά. Αντί για 160.000 ε, άτομα, τελείως αυθαίρετος αριθμός, αλλά τέλος πάντων, πετύχαμε να επανακαταστήσουμε περίπου 1000 Βέβαια, αυτό αποδεικνύει ούτως ή άλλως ότι η λογική υπεριασύλου στα κατημέλη πρέπει να είναι διαφορετική. Η δική μου ανησυχία στον επίπεδο της ομάδας μου και η προσωπική μου ανησυχία είναι το αν μπορούμε να ενδιαφερθούμε ώστε κάποια κάτι μέλη να μην μπορούν να αρνούνται όπως θέλουν ε, την αλληλεγγύη προς την Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν διαρκώς οι ίδιοι για τα πάντα και για πρώτη φορά ε, να ζητούμε ε, αλληλεγγύη από όλες τις χώρες σε επίπεδο υπήρου και να μας λένε οι χώρες όχι, εμείς δεν πληρώνουμε. Αυτό ισχύει και για τη μετανάστευση και για το άσυλο. Διότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που τα, οι αιτήσει ασύλου είναι τόσες πολλές και τόσο πολύ να επικεντρωθούν σε μερικούς γεωγραφικούς προορισμούς που να χρειαστεί να γίνει επανακατανομή επί της ουσίας. Εάν συνεχίσουμε λοιπόν να αποτυγχάνουμε όπως κάναμε την πρώτη φορά, ε, δεν θα πετύχουμε τίποτα προς την αξιοπιστία μας και ούτε θα πείσουμε την Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη. Το δεύτερο που θέλω να πω, κύριε Επίτροπε, δεν ήσασταν εδώ, αλλά ο κύριος Τίμερμανς και η κυρία Μογκερίνη μας παρουσίασαν την προηγούμενη φορά στην ε, Ολομέλεια τη νέα λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα της μετανάστευσης σε σχέση με τις εξωτερικέ μας σχέσεις. Είναι ένα θέμα φοβερά αμφιλεγόμενο. Αντί να επενδύουμε στις εγκατεστάσεις της Αφρικής όπως κάνει η Κίνα, θα πρέπει να στηρίζουμε περισσότερο τις χώρες της Αφρικής που τελικά φαίνεται να τις κάνουμε να γίνουν και αυτές μικρά οχυρά της Αφρικής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Και το λέω και σε εσά και προ όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όσοι είναι υπεύθυνοι για τι εξωτερικέ σχέσει, έστω και ατύπω, να τα ξανασκεφτείτε όλα αυτά. Διότι για τα αφρικανικά κράτη βλέπουμε τακτικέ διακυβέρνηση που είναι τελείω αμφισβητήσιμε, τρομερά αμφισβητήσιμε. Δεν θέλουμε απλώ να φυλάνε τα σύνορά μα και να μην κάνουμε τίποτα για την Αφρική. Και αυτό δεν θα προσφέρει τίποτα και σε εμά. Θα πρέπει εν τέλει η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν αναπτυχθεί η Ήπειρο τη Αφρική, με μέσα πολύ περισσότερα από ό,τι τώρα έχουμε προβλέψει, εάν δεν πετύχουμε να ε, παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την κατανομή των πόρων, πάλι θα αποτύχουμε. Σκεφτείτε για λίγο τι θα σήμαινε η Νιγηρία που τα 50 επόμενα χρόνια θα έχει 450 εκατομμύρια κατοίκους. Με μια σημαντική τρομοκρατική ομάδα στο βορρά της χώρας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη τη χώρα. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να, συμβαίνει, να σημαίνει αυτό προς την μετανάστευση. Πόσο θα μπορούσαμε να τη διαχειριστούμε. Και επειδή εξάλλησα το χρόνο μου, ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους ε, που έχουν ζητήσει το λόγο να, παρα... να προσπαθήσουν να περιοριστούν σε δύο λεπτά. Γιατί δεν θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε και δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο Αμπραμπόπουλο. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε κάποια λίγα ζητήματα. Μια πρώτη παρατήρηση. Τις τελευταίε εβδομάδε αναγνωρίσαμε πω η Τουρκία και πολλού πρόσφυγε, Αλλά δυστυχώ δεν μπορούμε να απευθύνουμε τον ίδιο έπαινο και σε όλα τα κράτη-μέλη μα Να πάρουν έστω και κάποιου πρόσφυγε. Και πιστεύω πω αν τα πράγματα παραμείνουν ω έχουν, δεν θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε αξιόπιστα με τρίτα κράτη και να τα πείσουμε να υποδεχτούν πρόσφυγε αν εμεί δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και πιστεύω πως τις επόμενες εβδομάδες πρέπει όσον αφορά το ζήτημα της μετεγκατάστασης να υπάρξει κάποια κινητικότητα. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία με την Τουρκία. Είχε σχεδιαστεί μια ανταλλαγή έναν προς έναν για κάθε σύρο που επιστρέφεται, υποδεχόμαστε έναν. Αλλά αυτό φυσικά δεν αφορά όλους όσους έρχονται μέσω Τουρκία στην Ελλάδα. Γιατί περιοριστήκαμε στην Συρία και δεύτερον, εάν όλοι οι πρόσφυγες που έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα επιστρέφονται, αυτό είναι συμβατό με το ατομικό δικαίωμα σε άσυλο αλλά και με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Και μία ερώτηση σχετικά με τις επερχόμενες κατευθυντήριες γραμμές περί ασύλου δεν είναι τόσο παλιές, δεν έχουν εκ, εκτελεστεί καν. Τώρα θα υπάρξουν νέες προτάσεις. Η ερώτησή μου, μπορείτε να διασφαλίσετε πως οι προτάσεις της Κομισιόν θα οδηγήσουν σε μία περαιτέρω εναρμόνιση, αλλά πως τα πρότυπα δεν θα μειωθούν. Και μια τελευταία παρατήρηση για την πολιτική θεωρήσεων και δύο για την αμοιβαιότητα θεωρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ τίθεται το ερώτημα, θέλουμε να άρουμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων, όντως, επειδή θα είχε έντονες οικονομικές συνέπειες. Το μήνυμα μου προς εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πάντα, ναι βέβαια θα ήταν πρόβλημα, αλλά η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά του γηπέδου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και παρακαλώ μιλήστε με την κυβέρνησή σας επιτέλους να υλοποιήσει αυτά που δεσμεύτηκε και να τηρήσει την αμοιβαιότητα θερεώσεων. Και ελπίζω η Κομισιόν ως προς αυτό να κρατήσει μια σταθερή θέση απέναντι στις ΗΠΑ και να φροντίσει να υπάρξει κάποια κινητικότητα έτσι ώστε να έχουμε αμοιβαιότητα. Ευχαριστούμε κύριο Σκύρχοπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ως συνήθως εκτιμούμε την προθυμία σας να έρχεστε στην Επιτροπή μα για να συζητούμε με τόσο ανοιχτό τρόπο. Είναι προφανέ για όλου μα το Κοινοβούλιο ότι οι αποφάσει που λαμβάνουμε τώρα είναι κρίσιμη σημασία για το μέλλον. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε περάσει τέτοιε δυσκολίε η Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την ασφάλειά τη και τη μετανάστευση. Επίτροπε, θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει με, ε, με κοινού πόρου και προσπάθειες και ελπίζω να μπορείτε να επαφίεστε στις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου και στις δυνάμεις μας που θα τις ενώσουμε με τις δικές σας και στο μέλλον. Στην πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου μιλήσαμε για τη λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μας και συμφώνησα και εγώ. Είναι μεγάλη σημασία για την ασφαλειά μα. Θα ήθελα αν μπορείτε να μα πείτε πόσο φιλόδοξου στόχου έχουμε ω προ αυτό και τι βήματα μπορούμε να περιμένουμε στο ερχόμενο χρονικό διάστημα. Ω εισηγητή για τον ερχόμενο φάκελο για το Eurodac και το Equis, θα ήθελα να βεβαιωθούμε ότι όλε οι βάσει δεδομένων ε, επικοινωνούν μεταξύ του και ότι όλα τα απαραίτητα νομικά εχέγγυα ε, προβλέπονται ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα αυτά απομονωμένα και ε, για την μετανάστευση τώρα. Ήθελα να ρωτήσω για τη Συμφωνία Επανεισδοχή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Μπορείτε να μα πείτε πότε μπορούμε να περιμένουμε την πρώτη έκθεση για το πώ λειτουργεί και αξιολόγηση για το πώ προχωρά ως τώρα η εφαρμογή της συμφωνία. Υπάρχει θετικό αντίκτυπο στον αριθμό των ε, ατόμων που επιστρέφονται και πώς ε, θα διαμορφωθούν στο μέλλον και τα για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα επιδιωχθούν οι στόχοι στο πρόγραμμα Ντεμέτε και είναι αυτό μια ε, μέθοδος να πιέσουμε περισσότερο τις τρίτες χώρες για επιστροφές και επανεισδοχές. Πόσο θα φανούν επιφαλεκτικές οι τρίτες χώρες ως προς αυτό και για τα θεμελιώδη δικαιώματα ή την ασφάλεια σε επιστροφή για επιστροφή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Πρέπει αυτά να λαμβάνονται πάντα ως κριτήρια υπόψη. Και να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι δεν ε, μπορούν να πάρουν διεθνή προστασία, οπότε πρέπει να επιστραφούν. Όμως πρέπει να σκεφτούμε αν είναι ασφαλεί εκεί που θα τους ξαναστείλουμε και να φροντίσουμε τους πλέον ευπαθείς εφόσον δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι ουρές για επιστροφή μεγαλώνουν. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πως θα στηρίξουμε και αυτέ τι χώρε και τι οικονομικέ ευθύνε αναλογούν και σε εκείνους για την αντιμετώπιση μια διεθνούς κρίσης. Δεν μπορούμε να ε, αναθέσουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες τη διαχείριση της δικής μας κρίσης, αλλά ούτε μπορούμε να τα αναλάβουμε όλα μόνοι μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο που ήρθε να περάσει το απόγευμα του μαζί μας. Είναι πάντα ενδιαφέρον να ανταλλάσσουμε ε, για θέματα μαζί σας και πραγματικά το εκτιμώ. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πώς θα συνεργαστούμε ε, με τρόπο ομαδικό, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την επίτευξη ενός καλού ψηφίσματος για το Δουβλίνο, για τις διαδικασίες, για την υποδοχή, για την ΕΑΣΟ. Είναι όλα τόσο στενά συνδεδεμένα που χρειάζεται αυτή η κοινή προσέγγιση για να προχωρήσουμε με ένα συνεκτικό τρόπο με όλα αυτά τα θέματα. Είχα μόλις μία συνάντηση με ΜΚΟ πέντε λεπτά πριν έρθω στην αίθουσα και μου είπαν, και δεν είναι η πρώτη φορά, ε, και μάλιστα εν χορό, πως έχουν σοβαρές ανησυχίες για το όσα κάνουμε εδώ, γιατί φοβούνται πως δημιουργεί ένα σύστημα το οποίο ε, ουσιαστικά προσογγίζει την προσέγγιση της Αυστραλίας. Είναι μια προσπάθεια να τους σπρώξουμε μακριά. Ξέρω πως έχετε εσείς τις καλύτερες προθέσεις και εμείς το ίδιο και αυτό έχει ήδη υποθεί ε, στα πλαίσια της έκθεσης για την ολιστική αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Όμως, όταν ακούμε τέτοιου είδους ανησυχητικά μηνύματα και όταν ακούμε τις δηλώσεις των υπουργών που μας δημιουργούν ανησυχία στα κράτη-μέλη που θέλουν τη συμφωνία αυτή με την Τουρκία, θέλουν να την επαναλάβουν ε, με τη Λιβύη για παράδειγμα. Ο υπουργό της Σουηδίας για τα ευρωπαϊκά θέματα το είπε τις προάλλες, το είπε ο ε, Αυστριακός Υπουργός Εσωτερικών. Αυτά τα μηνύματα είναι ανησυχητικά και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Πρόκειται να επεκτείνουμε αυτή την τακτική που είναι να σπρώχνουμε τα εξωτερικά κάμας μας ε, σύνορα προς τις ε, τρίτες χώρες και να απαρνηθούμε τις ευθύνες που έχουμε στην Ευρώπη για ανθρώπους που υποφέρουν. Επίσης, για την μία αμοιβαιότητα στο θέμα των θεωρήσεων με τις ΕΠΑ Πρόσφατα ε, εστάλει μια επιστολή και νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς ποια είναι η νομική υποχρέωση που απορρέει από το θέμα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ θετικό σήμερα το απόγευμα να γνωρίζουμε από εσάς ή να μας επιβεβαιώσετε πως ε, θα λάβουμε μια κατεξουσιοδότηση πράξη για το συγκεκριμένο θέμα της αμοιβαιότητας της θεωρήσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μάθω για τα εξή κάτι περισσότερο. Για τη συμφωνία με την Τουρκία. Κοιτάξαμε ακριβώ την κατάσταση σε Ελλάδα και Τουρκία και έχω τι εξή ερωτήσει. Όλα τα μέτρα και υποστήριξη που έχουν υποσχεθεί στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν. Αυτό αφορά τους εμπειρογνώμενες, την υποστήριξη, στην επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου. Όλα αυτά έχουν γίνει ναι ή όχι. Και ποια η θέση σας όσον αφορά την κριτική πολλών προσφύγων. Ότι παραδείγματο χάρη αίτηση ασύλου επεξεργάζονται ή πρόκειται να επεξεργαστούν μέσω Skype, το οποίο αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για πολλού. Όσον αφορά τη συμφωνία με την Τουρκία, διαπιστώσαμε ότι πολλοί δεν μπόρεσαν καν να αιτηθούν άσυλο ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Είχαμε περιπτώσει όπω διεμφυλικών ανθρώπων που βρήκαμε στην Τουρκία σε φυλακές Απέλαση και μάλιστα απέλασης προς το Ιράν, ένα σκάνδαλο. Βρήκαμε Πακιστανούς, οι οποίοι δεν πρόκειται να, να γίνουν δεκτοί στις χώρες προέλευσής τους. Έχουμε αφγανικές οικογένειες, στις οποίες δεν επιτραπεί και η οικογενειακή επανένωση. Έχουμε δηλαδή μία μη επεξεργασία αιτήσεων ασύλου και ιδίω εάν πρόκειται για μη σύρου. Σχετικά με αυτό θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα. Το δεύτερο, η απελευθέρωση των θεωρήσεων με την Τουρκία. Όλα αυτά έχουν παγώσει. Έχουμε κάποια νέα. Η Κομισιόν θα παραμείνει στη θέση τη ότι δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτω τίποτα όσον αφορά το ζήτημα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων και την τήρηση των 72 κριτηρίων. Όσον αφορά το Δουβλίνο, μία και μόνο ερώτηση ο λεγόμενος μηχανισμός δικαιοσύνης, η διόρθωσης. Πόσα κράτη-μέλη θέλουν να υποστηρίξουν επί του παρόντος ένα τέτοιο διορθωτικό μηχανισμό. Και το δεύτερο, η καταπολέμηση των διακινητών. Λέγεται συνέχεια πως πρέπει να καταπολεμήσουμε περισσότερο τους διακινητές και να διευρύνουμε την καταπολέμηση. Τι πέραν των μέτρων που προβλήθηκαν ήδη για την Frontex πρόκειται να υπάρξει, τι καινούριο πρόκειται, τι ποιοτικά καινούριο πρόκειται να προσταθεί σε αυτό. Η κυρία Φεράρα, η κυρία Σκάλου συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω για την Ελλάδα υπήρξαν αναφορές. Η Προεδρία, η Ολλανδική Προεδρία είπε πως δεν είναι ευχαριστημένη με τις αποφάσεις, τις δευτεροβάθμιες αποφάσεις ασύλου στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές βέβαια μπορεί να μην είναι όπως τις περιμένουν κάποιοι άλλοι, αλλά οι επιτροπές ασύλου υπάρχουν εκεί για να λαμβάνουν αποφάσεις. Δεν ξέρω αν είχατε στο Συμβούλιο κάποια συζήτηση γι' αυτό και μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πώς πήγε, τι αντιδράσει υπήρξαν. Επίσης υπήρξαν καταγγελίες από δικηγόρους πως η Άσο απορρίπτει αγωγές από άσυλο, δηλαδή ότι έχουμε μια απόρριψη κατά 100% και πως η αιτιολόγηση δεν γίνεται σωστά. Διερευνάει η Κομισιόν κάτι τέτοιο. Επίσης σήμερα υπάρχει το ζήτημα να επιστρέψει η Ελλάδα στο σύστημα Δουβλίνου έως το τέλος του χρόνου. Θα αξιολογούσατε την κατάσταση κατά έναν τρόπο ώστε έως το τέλος του έτους θα έχουμε αποδεκτές εγκαταστάσεις υποδοχής χωρίς υπερπληθυσμό από ετούντες άσυλο. Πιστεύω είναι μια αισιόδοξη προσέγγιση. Και από ό,τι φαίνεται η Άσο συνέταξε μια έκθεση σύμφωνα με την οποία η Τουρκία δεν είναι ικανή να επεξεργαστεί αιτήσεις ασύλου και λέγεται πως αυτή η έκθεση δεν δημοσιεύτηκε λόγω του πολιτικά αμφιλογόμενου περιεχομένου της. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτή την έκθεση παρακαλώ. Επίσης προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτή τη διασυνοριακή συνεργασία με τρίτες χώρες. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης ασχολούμαστε επίσης με αυτό. Αυτό σημαίνει συνήθως την αποστολή εξοπλισμού, την εκπαίδευση συνοριοφυλάκων, έτσι ώστε να υπάρχει μικρότερη διέλευση προσώπων από τα σύνορα. Αλλά ποια είναι, ποιον, ποια είναι ακριβώς η διαχείριση σύνορων που γίνεται. Η κυρία Φεράρα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε Αβραμόπουλε. Και εγώ θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα η αναθεώρηση του συστήματος ασύλου, ιδίως ο κανονισμός του Δουβλίνου. Τώρα πλέον τα λέμε σε κάθε ευκαιρία, στην Επιτροπή Λίμπε, στην Ολομέλεια. Είναι μια πρόταση, μια πρόταση αναθεώρησης που δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει γιατί συνεχίζει να τιμωρεί τι πρώτε χώρε, τι ίδιε χώρε, τι πρώτε χώρε, τι πρώτη εισόδου λόγω τη γεωγραφική του θέση. Με ένα διορθωτικό μηχανισμό, ο οποίο ε, ουσιαστικά δεν είναι προ ε, είναι απλώ αντιδρά, δεν ε, προλαμβάνει. Όπω το είπε και η Επιτροπή Λίμπε με μια μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό μας και όπως είπε και η Άσο θα πρέπει να μην λειτουργεί μόνο για την επανακατανομή των ανθρώπων αλλά κάπως να προλαμβάνει και τις χώρες πρώτης εισόδου. Η χώρα πρώτης εισόδου καθίσταται τελικά υπεύθυνη ακόμη και αν ο μετανάστης δεν έχει δικαίωμα στη διεθνή προστασία. Επιστρέφει στη χώρα προέλευσης και μετά επιστρέφει δεύτερη φορά στην Ευρώπη. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα αυτό που δεν λειτουργήσε ως τώρα θα συνεχίσει να είναι κάτι που και στη νέα πρόταση θα μας προβληματίζει. Λίγα κράτη-μέλη όμως επηρεάζονται από αυτό. Η πραγματική κατανομή, ε, η ίση κατανομή των ευθυνών δεν έχει ακόμη υπάρξει όπως ζητά το άρθρο 80 της συνθήκης. Γι' αυτό λοιπόν ε, έχω να ρωτήσω ε, η βούληση όπως εκφράστηκε και από το Κοινοβούλιο στην ε, εγκεκριμένη από το Κοινοβούλιο έκθεση για την ολιστική προσέγγιση στη Μεσόγειο. Πώς θα ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, η συμφωνία με την Τουρκία. Και εδώ είμαστε πολύ επικριτικοί στη στάση μας Με μια συμφωνία που δεν είναι διεθνή συμφωνία, δεν είναι σύμφωνο, αλλά ήταν απλώ μια δήλωση, μια πολιτική δήλωση. Δεν έχουμε καμία διασφάλιση ότι η Τουρκία από την πλευρά τη θα σεβαστεί τι υποχρεώσει που ανέλαβε. Αυτή τη στιγμή ε, έχει υποτίθεται να λάβει κάποιε υποχρεώσει, δεσμευτικέ μάλιστα. Ε, θα ακολουθηθούν κάποιε τακτικέ νομοθετικέ διαδικασίε, όπω η απελευθέρωση των καθεστώτων καθεωρήσεων ή ε, ο αντίκτυπο των προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν με κάτι που απλώ θα καθησυχάσει και θα διασφαλίσει την Τουρκία με δική μα δέσμευση, από την άλλη δεν εξισταθμίζεται, δεν αντισταθμίζεται αντισταθμίζεται με μια άλλη κίνηση από την Τουρκία πέρα από μια πολιτική γενικώ δήλωση. Από την Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε ω προ την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ελευθεροτυπία. Είναι δύσκολο να την χαρακτηρίσουμε ασφαλή χώρα. Ακόμη δεν έχει κυρώσει την σύμβαση τη Γενέβη για του πρόσφυγες του 1951. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Τουρκία θα σεβαστεί τα δικαιώματα των μεταναστών, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαβεβαίωση ούτε τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τελευταίο σχόλιο για το Migration Compact, το σύμφωνο αυτό για την μετανάστευση. Έχετε σκεφτεί ένα μη σύστημα παρακολούθησης για την αναβήμα και σε κάθε λεπτομέρεια χρήση των κοντιλίων, διότι ακόμη χώρε με, ε, με απολυταρχικά καθεστώτα, με τάσει ε, καταστολή και καταπίεση πιστεύω ότι τα κοντήλια θα φέρουν στα χέρια του. Δεν θα πάνε προ την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Έχει προβλεφθεί μια, μια δράση παρακολούθηση, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε ακριβώ πώ θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και τι είδου αποτελέσματα αναμένουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χολμάγκερ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο ε, τι συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ε, να σας πω πως 1.300 ε, ετούντες άσυλου ψάρεψαν από τη θάλασσα κοντά στις ακτές της Ιταλίας. Και έχετε ακούσει ποιε είναι οι προτάσει αυτή τη στιγμή για να ε, απελευθερωθεί το καθεστώς χορήγησης ε, για το Κωσυφοπαίδιο, για την Τουρκία, για την Ουκρανία, για τη Γεωργία όλο και περισσότερο ε, μετανάστευση, μαζική μετανάστευση από τις χώρες αυτές. Σας παρακαλώ, μην μας δίνετε την εντύπωση ότι οι κάτω χώρες έχουν ανάγκη από περισσότερους ετούντε εργασία, γιατί εμάς τα επίπεδα ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλά και επίσης το εργατικό μας ε, δυναμικό είναι πάρα πολύ έντονο και αυτή τη στιγμή τους δίνουμε το λαχείο για να έρθουν όλο και περισσότεροι μετανάστες, με όλες τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό και ξέρετε τι ζημιά έχει υποστεί η κοινωνία μας όλα αυτά τα φαινόμενα. Και δεύτερον, έχετε το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση το οποίο έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατάσταση στις χώρες μας και στις πόλεις μας έχει δείξει πως η ενσωμάτωση των ετούντων άσυλο τους έχει δώσει μεν δικαιώματα, αλλά δεν τους έχει επιβάλει οποιαδήποτε υποχρέωση. Και πιστεύω πως θα έπρεπε να τους στείλουμε πίσω στη χώρα τους η ενσωμάτωση δεν λειτουργήσε. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως τα άτομα αυτά προσαρμόζονται στους δικούς μας κανόνες, στους δικούς μας νόμους και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, στα πλαίσια του ρόλου που παίζει και το Ισλάμ. Γιατί ξέρετε πως είχαμε και επεισόδια για τα οποία η Κομισιόν απλώς έκλεισε τα μάτια. Λοιπόν, οι προτάσεις αυτές κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αφαιρεθούν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Uh, και τώρα Ολοκληρώνουμε με τους συντονιστές και θα δώσω και πάλι το λόγο στον Επίτροπο. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, κάποιον ξέχασα. Θα ήθελα τουλάχιστον να κρατήσω αποστάσεις από αυτή την άποψη που ακούστηκε από το πώς χαρακτηρίστηκαν ως τυχοδιώκτες οι πρόσφυγες. Θεωρώ πως χαρακτηριστηκαν ως τυχοδιοκταση είναι απέσιο αυτό που είπε η προαλήσασα. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Παρακαλώ, έχετε κατά ότι έχουμε 14 άλλα μέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια παρατήρηση. Πολλοί από σας θέσατε και πάλι ένα πολύ ευαίσθητο ερώτημα στο ένα ζήτημα της αλληλεγγύης συμφωνούμε ως προς αυτό και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως το έχουμε συνέχεια κατά νου. Πως πρέπει να το δείχνουμε και πρακτικά. Επειδή η αλληλεγγύη και η ευθύνη είναι ωραίες λέξεις αλλά δεν είναι συνθήματα. δεν πρόκειται για ηθικές αξίες, αλλά επίσης νομικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται ρητό στις συνθήκες. Εμεί θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το μερίδιο τη ευθύνη που του αναλογεί όσον αφορά την μετεκατάσταση. Τι τελευταίες εβδομάδε είδαμε, όπω είπα και πιο πριν, κάποιε θετικέ εξελίξει. Προ το παρόν έχουμε κάποια κινητικότητα. Αργή, αλλά σταθερή. Τώρα είναι η στιγμή να επισπεύσουμε. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας με μια αίσθηση ευθύνης και αλληλεγγύης. Λοιπόν, κυρία Ζήπελ, δείξατε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις όσον αφορά την Τουρκία. Στην Τουρκία οι Σύριοι μπορούν να καταχωρηθούν για ένα προσωρινό καθεστώς. Οι μη Σύριοι μπορούν να ζητήσουν διεθνή προστασία, επικουρική ή υπόρρος προστασία. έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα από την τουρκική πλευρά πως η Τουρκία δεσμεύεται να δεχτεί νέες αιτήσεις ασύλου εντός έξι μηνών από τη συμφωνία και να επεξεργαστεί τη συμφόρηση αιτήσεων. Το ζήτημα είναι να μην θέσουμε την προτεραιότητα στην ταχύτητα και όχι στην ποιότητα της επεξεργασίας των αιτήσεων. Ναι, η Τουρκία έκανε βήματα για να βελτιώσει την πραγματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση για τους Σύρους και για τους μη Σύρους. Και μιλώ για μια εκπαίδευση η οποία παρέχεται δωρεάν για όλους τους Σύρους και φυσικά τους μη Σύρους που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας. Καθώς μιλούμε για την Τουρκία, θα ήθελα να σας πω πως η επιτυχία της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας είναι μια κοινή δήλωση, δεν είναι μια συμφωνία. Γνωρίζετε τη διαφορά όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, αλλά είναι μια δέσμευση. Η επιτυχής εκτέλεση της δήλωσης αυτής είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας, για την Επιτροπή και συνεχίζουμε να κάνουμε το παν δυνατόν για να παρέχουμε υποστήριξη και ειδικευμένη γνώση στις ελληνικές και τουρκικές αρχές. Η δήλωση αυτή έχει ήδη αποτελέσματα. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Έχουμε μία οξιαμείωση των αριθμών των μεταναστών που περνούν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Υπάρχει το γεγονό ότι περισσότεροι από 400 μετανάστε επιστράφηκαν στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων 31 Σύρων, οι οποίοι επέστρεψαν εθελοντικά και πως πάνω από 300 Σύριοι μετεγκατασταθήκαν από την Τουρκία. Όλα αυτά αποτελούν αποδεκτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δήλωσης. Δεν είναι κάτι το θεαματικό, αλλά δείχνει πως άρχισε να λειτουργεί. Έχουμε βέβαια ακόμα προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως την αύξηση των ικανοτήτων των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο έγκαιρα και αποτελεσματικά. Όσον αφορά την αμοιβαιότητα θεωρήσεων, η κυρία Ζήπλο ρώτησε κάτι. Η Επιτροπή εξέφρασε στην Επιτροπή του κυρίου Μοράλες πως λαμβάνει γνώση του ζητήματος. Το προτίθεται το Κοινοβούλιο να προβεί σε ψήφισμα για το ζήτημα. Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν από το κολέγιο. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας ενημερώσω για τη χρονική στιγμή. Όσον αφορά την ανακοίνωση της 10 η Απριλίου, η ε, Κομισιόν θεώρησε κατάλληλο να παρουσιάσει μια εξήγηση του πιθανού αντικτύπου της αμοιβαιότητας των, της άρσης της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων. Θέλουμε επίσης να αρχίσουμε έναν διάλογο με περιεχόμενο πριν προβούμε σε βήματα τα οποία μπορεί να έχουν αντίθετες και αρνητικές συνέπειες. Μετά τη συνεδρίαση του Λίμπεν με τις αφρικανικές με τους αφρικανικούς φορείς πιστεύω πως η προσέγγιση αυτή είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και επίγουσα. για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της εποχιακής άφηξης μεταναστών και προσφύγων στην Κεντρική Μεσόγειο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επί χρόνια. Αλλά φυσικά ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα βρίσκεται στο επίκεντρο της εφαρμογής. Οι ροές αυτές προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική και φτάνουν σε εμά κάθε χρόνο. Εκμεταλλευόμενοι τη διαπερατότητα των συνόρων αφρικανικών κρατών. Παρελπτόντως, θα ήθελα να σας αναφέρω την διαφορά μεταξύ αυτού που έχουμε κάνει με την Τουρκία και αυτού που γίνεται εδώ. Η Τουρκία είναι εταίρος μας, συνομιλητής μας, και συνεργαζόμαστε με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο μπορεί να γίνει με τη Λιβύη. Η Λιβύη δυστυχώ ακόμη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Είναι ένα αποτυχημένο κράτο. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε ένα συνομιλητή και εκεί. Όταν έρθει η στιγμή, αυτό που θα κάνουμε δεν θα είναι μια συμφωνία αντίγραφο, copy-paste, αυτό που κάναμε με την Τουρκία. Θα έχουμε λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε χώρας. Ενώ οι αφήξει από την Αίγυπτο διπλασιάστηκαν, η μεγάλη πλειοψηφία των παράτυπων μεταναστών από την υποσαχάριο Αφρική και όλη την Βόρειο Αφρική συνεχίζει να ξεκινάει το ταξίδι του από τη Λιβύη Γι' αυτό και πρέπει επιγόντως να εμπλέξουμε τις χώρες προέλευσης των ροών αυτών και να τις πείσουμε να συνεργαστούν μαζί μας. Και επίσης να πείσουμε τις χώρες τρανζιτ, διέλευσης να συνεργαστούν για την αποτροπή του φαινομένου αυτού. Αναφέρομαι σε 7 έως 8 χώρες της περιοχής αυτής και πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς στις συνομιλίες μαζί τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η ανάπτυξη είναι πρώτη προτεραιότητα δική μας. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές. Το κάνουμε επί δεκαετίες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά από την πλευρά τους πρέπει πάντοτε να δείχνουν περισσότερη ευθύνη και να ανταποκρίνονται θετικά στις συμφωνίες μας για να σταματήσει η παράτυπη μετανάστευση. Και φυσικά πρέπει να τους πείσουμε να δεχτούν τους υπηκόους τους. Υπάρχουν και χώρες που, στις οποίες κατοικούν μεγάλες κοινότητες μεταναστών, οι οποίες πρέπει να προστατεύσουν καλύτερα τα δικαιώματα των μεταναστών για να αποφύγουμε και δευτερογενείς ροές. Πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους αντί να αρχίσουν το επικίνδυνο αυτό το ταξίδι. Οι υπήκοοι των χωρών αυτών μπορούν στις χώρες τους να κτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ζωές τους. Όσον αφορά τις συνδίκες υποδοχής στην Ελλάδα, η Κομισιόν συνεργάζονται πολύ στενά με τις ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση του ζητήματος και τα κέντρα καταγραφής hot spots στην Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμμο είναι πλέον πλήρως λειτουργικά επί των παρόντων προσαρμόζονται στον στόχο της πραγματοποίησης επανεισδοχών στην Τουρκία. Όπως λέω, η συμφωνία εφαρμόζεται ήδη. Το αυστραλιανό μοντέλο το αυστραλιανό, μοντέλο δεν είναι το πρότυπό μας γι' αυτό. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις. Κάτι είπε και με ρώτησε η Σκα Κέλλερ. Υπό το πρίσμα της συμφωνίας αυτής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας όλες οι αιτήσεις ασύλου γίνονται κείμενο δεξεργασίας αναπερίπτωση. Και σίγουρα δεν υπάρχουν αυτόματες επανειδοχές ούτε έντυπα μπλάνκο. εξετάζουμε κάθε περίπτωση, κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Οι αποφάσεις δεν σημαίνουν κατά ανάγκη πως οι αιτήσει για άσυλο θα εξετάζονται όπως το αναμένουμε. Γνωρίζετε πως η σύσταση των Επιτροπών Ασύλου είναι κυρίαρχη αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές, όπως γνωρίζετε, δημιουργήθηκαν υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες πριν από μερικά χρόνια και για διαφορετικούς σκοπούς. Οι παλιές επιτροπές αντικαθίστανται τώρα και θα συνεχίσουν και θα υπάρξει μια νέα νομοθεσία στην Ελλάδα η οποία θα διασφαλίσει την νομιμότητα, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών αρχών. Εδώ και πέντε χρόνια έχουν σταματήσει οι μεταφορές Δουβλίνου. είδαμε ότι παξιμιώθηκε πολύ πρόοδος. Αλλά γενικά η κατάσταση όσον αφορά το συντούς άσυλο είναι ακόμα ανεπαρκής και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες μέχρι έως ότου η Ελλάδα να μπορέσει να ξαναπροβεί σε μεταφορές του Δουβλίνου. Οι εγκαταστάσεις, κατάλληλες συνθήκες ζωής για όλους τους ετούντες, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο των ελληνικών αρχών και τον Σεπτέμβριο θα προβεί μια έκθεση. Έχουμε το στόχο να, δημα... να διπλασιάσουμε τις μεταφορές Δουβλίνου έως το, 2010... έως το φθινόπωρο του 2016. Θα δούμε κατά πόσον η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη έως τότε. Θα σταματήσω τώρα και θα επανέλθω αργότερα για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Γκικόμπε, έχω κάτι για σας. η προτεραιότητά μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να επαναλάβω για μία φορά ακόμα πως προσπαθούμε πολύ να πείσουμε όλα τα κράτη-μέλη να εμπιστευτούν περισσότερο το ένα το άλλο, το άλλο και να αρχίσουν μια γενική συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και πληροφοριών μυστικών υπηρεσιών. Και πρέπει να είμαι ειλικρινή. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένο με την κατάσταση. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και για την πρόσφατη νομοθεσία περί τρομοκρατίας και πυροβόλων όπλων. Και εν ώψη της απειλής αυτής η νομοθεσία είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως το αντιτρομοκρατικό κέντρο της Europol είναι πλήρω λειτουργικό πλέον και πως οι οργανισμοί πρέπει να συνεργάζονται μαζί, μεταξύ του. Ο θεσμός αυτός πρέπει να ενισχυθεί καθώς και οι αρχές επιβολής του νόμου για την ανάλυση του, της τρομοκρατίας και απειλών έτσι ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση και πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου η θέση μου σήμερα το απόγευμα, αλλά 16 ε, συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα επιτρέψω σε όλους να τον λάβουν, όμως θα έχετε ένα λεπτό ο καθένας. Εάν όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε τις απαντήσεις. Να προτείνω κάτι. Είμαι από του επιτρόπου που μου αρέσει πολύ να έρχομαι εδώ. Αλλά για να γίνει η συνεργασία μα λίγο πιο παραγωγική, ε, θεωρώ καλύτερα θα ήταν οι συζητήσει μα να πάρουν μια θεματική οργάνωση. Δηλαδή να μπορώ να δίνω μια συνολικότερη απάντηση, διότι πηγαίνω ερχόμαστε και επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Και πιστεύω ότι αυτό θα ε, συμβεί και τώρα στη συζήτησή μα. Είναι μια πρόταση, αν θέλετε να βρείτε ένα καλύτερο τρόπο κάπω για να οργανώνουμε τι παρεμβάσει. Το καταγράφουμε αυτό που είπατε, άλλη φορά ίσως, αλλά τώρα θα ζητήσω τους συναδέλφους να ε, βιαστούν και να μείνουν στο ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Κοέλιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ε, με ένα λεπτό προτιμώ να μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε και συγχαρητήρια για την ε, νυφαλιότητα με την οποία αναλάβατε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα, αυτό το φάκελο. Θέλω να κάνω τρεις πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, την ε, ε, επαναγκατάσταση και την απόκριση έκταξης ανάγκης. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα. Η Πορτογαλία είναι η δεύτερη χώρα σε απόκριση αιτήσεων ασύλου από την Ιταλία και από την Ελλάδα. Αλλά Έχουμε καταφέρει να επανακαταστήσουμε 2.200 άτομα μόλις. Συνεχίζουμε να αποτυγχάνουμε. Δεύτερη ερώτηση. Σε σχέση με όσα υπόθηκαν για την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια, μιλήσατε για την ε, μεταγκατάσταση, ε, για ένα μηχανισμό που θα ε, λειτουργεί εσωτερικώ, υποτίθεται, αλλά ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Θεματολόγιο για την Μετανάστευση πρότεινε τη δημιουργία ενό ε, πολυδύναμου κέντρου στο ε, Νίγηρα, αλλά τι πρόταση χρηματοδότηση υπάρχει εδώ. 4% των κονδυλίων που χρειάζονται για τη στήριξη τη Αφρική, έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη σωστά. Θα προταθεί κάτι από την Επιτροπή για τι χώρε προέλευση και διέλευση. Διότι πρέπει να προσέξουμε μην στοιχηματίσουμε πάλι στο λάθος άλογο στην κούρσα αυτή. Ευχαριστούμε και πάλι η κυρία Γκυγιόμ. Στα γαλλικά. Ε, θα αλλάξω θέμα. Ε, θέλω την άποψή σας για δύο θέματα. Ακούσαμε ότι θέλετε να ισχύει η γαλάζια κάρτα που είναι κάτι που ισχύει για τα υψηλών προσόντων προφίλ, αλλά ξέρουμε ότι πολλά είναι τα επαγγέλματα που στα διάφορα κάτι ακόμα δεν έχουν πετύχει αυτή την κατηγορία. Ε, τι θα γίνει λοιπόν για να συνδυαστούν αυτές οι δύο διαστάσεις και έπειτα για την ένταξη. 100.000 άτομα έχουν ζητήσει εθνικότητα από κάποιο κράτο μέλο τη μια την άλλη χρονιά. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι απόλυτο αριθμό ε, και κριτήριο το κατά πόσο ζητήθηκε η εθνικότητα ενό κράτου μέλου, η υπηκότητα. Όμω το ερώτημα είναι τι θα γίνει και με τη μετανάστευση ω προ αυτό. Ε, το πρόβλημα εμένει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρείται πλέον ως ένας ελκυστικός προορισμός. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα. Η κυρία Ριβονταλόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Τρει ερωτήσει για την νέα εταιρική σχέση με τι τρίτε χώρε. Με τι συγκεκριμένα μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία τη με τη Λιβύη. Η επιτυχία αυτή τη νέα εταιρική σχέση θα εξαρτηθεί από την οικονομική συμμετοχή των κρατών μελών, όπω και πολλά συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τομέα. Πώ τα κρατη υποδέχτηκαν την πρόταση αυτή και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη ε, θα ανταποκριθούν στις εκκλήσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρξουν ε, μέτρα πρότωσης κινήτρων για τις εμπορικές πολιτικές και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ε, παροτρύνουμε τις διάφορες χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε θέματα μετανάστευσης και εξέτασης ε, αιτήσεων ασύλου για όσους αρνούνται. Αυτό πώς θα γίνει συγκεκριμένα και πώς θα δοθούν ε, οικονομικές βοήθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις τρίτες χώρες για θέματα μετανάστευσης. Η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, για δύο θέματα που έθιξε ο Επίτροπο, η νέα προσέγγιση τη Ευρώπη για την εταιρική σχέση με τι τρίτε χώρε, ναι στην διπλωματία τη μετανάστευση, πλήρη στήριξη από εμά και επίση για την ένδοαφρικανική κινητικότητα. Πρέπει να είναι μια σωματική πτυχή αυτή τη νέα προσέγγιση και για τι θεωρήσει, σαφέ μήνυμα, να γίνονται σεβαστά όλα τα κριτήρια και κυρίω στήριξη προ του πολίτε. Δύο ερωτήσει για τη γαλάζια κάρτα. Αναμφισβήτητα, η αναθεώρηση που μα προτάθηκε, η ανακοίνωση τέλο πάντων, είναι ένα βήμα πρόοδου. Όμω γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δύο δυσκολίε παραμένουν. Πρώτον, η διαφορά μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών των 28 κρατών μελών και από την άλλη η έλλειψη ε, προθυμία από τα κράτη-μέλη για να προωθήσουν τη γαλάζια κάρτα. Σε εθνικό επίπεδο ξέρουμε ότι πολλά κράτη σε ό,τι αφορά την εθνική του νομοθεσία έχουν του ίδιου στόχου με τη γαλάζια κάρτα. Μεν, αλλά πολύ συχνά επιχειρηματίε ε, ανατρέχουν σε αυτού του εθνικού στόχου. Οπότε παραμένει το ερώτημα πώ μπορούμε να κάνουμε κάτι από κοινού για να προάγουμε αυτό το ευρωπαϊκό εργαλείο. Ένα εργαλείο που θα κάνει την Ευρώπη πιο ελκυστική. Είναι ένα εργαλείο κλειδί για τη μεταναστευτική μα πολιτική και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια σαφέστατη απάντηση σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε κυρία Γκαμπρίλη, κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ένα λεπτό είναι πραγματικά πολύ πολύ λίγο. Αλλά θέλω σε κάθε περίπτωση να σας ευχαριστήσω για την ε, συστηματική σας παρουσία εδώ και για τη δουλειά σας στην Επιτροπή. Πραγματικά συμμερίζομαι μαζί σας την παρατήρηση ότι πραγματικά δυστυχώς η μετανάστευση γίνεται ένα φαινόμενο που αποδεικνύει την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Και ενώ αληθεύει πρέπει να προσπαθήσουμε για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, πραγματικά χρειάζεται μια στρατηγική μακροπρόθεσμη, η οποία να προβλέπει παρεμβάσει πραγματικά αποτελεσματικέ. Κατά την άποψή μου, αυτό θα ήταν ένα κίνητρο και θα ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά σε αυτό το τομέα. Ε, δύο ερωτήσει τώρα. Ε, η πρώτη. Γνωρίζουμε καλά ότι πέραν των δραματικών συνθήκων των χωρών προέλευση των μεταναστών, Αυτό ε, προκαλεί διακίνηση, εμπορία ανθρώπων και φυσικά το μεταναστευτικό φαινόμενο. Έχουν γίνει λίγα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν γίνει, πιστεύετε, αρκετά από την ε, Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε την διακίνηση, την εμπορία μεταναστών. Αυτού που είναι διακινητέ και κερδίζουν από αυτήν την ε, ιστορία. Και επίση ω προ το σύστημα ασύλου. Σίγουρα είναι θετικό βήμα το, η στήριξη τη Eurodac και η ASO ω Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο. Όμω, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του συστήματο του Δουβλίνου δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους ενδιασμούς που εξέφρασαν εδώ τόσοι συνάδελφοι, ιδίω ο συνάδελφο Φεράρα. Πραγματικά μου φαίνεται ότι μεταξύ των πιθανών λύσεων για να αναθεωρηθεί το σύστημα του Δουβλίνου, μάλλον επελέγει η λύση που είναι λιγότερο φιλόδοξη. Αφήνει κι άλλη μια φορά τα κράτη-μέλη πρώτη άφηξη, αφήνει σε αυτού την ευθύνη να αντιμετωπίσουν όλε τι δυσκολίε. Οπότε δεν επιλύει με πραγματικά δραστικέ λύσει το όλο θέμα. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Κύριε Επίτροπε, θα συμφωνήσω και εγώ με τα όσα σας ζήτησε ο κύριος Κουέγιο. Γιατί δεν λειτουργεί για την Πορτογαλία το σύστημα. Γιατί πήγατε και η Πορτογαλία δηλώνει συνέχεια πως είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη να υποδεχθεί κόσμο. Τόσο λίγοι έφτασαν σε εμά. Το είπατε κι εσείς άλλωστε. Το σύστημα των hot spot είναι έτοιμο. Μπορεί να εφαρμόσει τη συμφωνία με την Τουρκία και παρόλα αυτά δεν είναι έτοιμο να εξετάζει ε, εξατομικευμένα τις αιτήσει ασύλου ε, για να φύγει αυτός ο κόσμος για την Ευρώπη. Και για το λόγο αυτό δεν έρθε κανείς από τα hot spot ούτε στην Πορτογαλία ούτε κάπου αλλού. Εντάξει. Για τη Λιβύη έχετε απόλυτα δίκιο, δεν υπάρχει εταίρος που είναι τον οποίο να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε. Όμως αυτό που διπλασιάζεται είναι οι ζωέ από την Αίγυπτο και αυτό έχει μια άμεση σχέση με τη Συρία, όχι μόνο με, μετοχ... με εποχιακές μετακινήσεις από την Αφρική. Επίση, η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσπαθεί να αποδείξει πόσο πόσο καλά πάει η συμφωνία με την Τουρκία και είναι σε άρνηση για το θέμα της Αιγύπτου. Και αυτή τη στιγμή με την Αιθιοπία έχουμε μια χώρα η οποία σκοτώνει τους πολίτες της, που είναι απολύτως μη δημοκρατική, που δημιουργεί πρόσφυγες και μετανάστες και έχετε μαζί τη συμφωνία. Ε, σήμερα προσπαθήσατε να εξασφαλίσετε ότι υπάρχουν ασφαλείς και νόμιμες οδοί έτσι ώστε να μην δρουν τα δίκτυα. Θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της συμφωνίας ή αυτή η συμφωνία απλώς κάνει υποεργολαβική ανάθεση εξωτερική του προβλήματος. Η κυρία Ιντβαλτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στα γρήγορα, Επίτροπε, εσείς δεν απαντήσατε στην ερώτηση της συναδέλφου μου ή της κυρίας Βίκστρομ γιατί δεν προτείνεται κατεξουσιοδότηση πράξη για την αμοιβαιότητα στον χώρο των θεωρήσεων. Όσα απαιτείται και δεύτερον για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, μιλήσαμε για την διαλειτουργικότητα των τεχνικών δεδομένων στις βάσεις, αλλά αυτό είναι τεχνικό θέμα και δεν ξεπερνιέται έτσι ο δισταγμός των κρατών πολλές φορές, για να μην σας πω η απόλυτη άρνηση να μοιραστούν πληροφορίες, που αποτελεί πολιτικό πρόβλημα. Εσείς τι θα προτείνετε, υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Και επίσης, εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο πολύ συχνά ζητάμε μία σε βάθος ανα, αξιολόγηση του toolkit για τα αντιτρομοκρατία. Γιατί βλέπω ότι χάνει ε, και χάνει Και κάνουμε πάρα πολλά, διαθέτουμε πόρους και το μόνο που κάνουμε είναι να αυξάνουμε το επίπεδο ανασφάλειας γύρω μας. Και το τελευταίο που έχω να πω, δεν μοιάζουμε να καταλαβαίνουμε το φαινόμενο με τον τρόπο που η σφαγή αμέσως ε, το Ορλάντο θεωρήθηκε ως ε, ε, Ισλαμική τρομοκρατία και τώρα που βγαίνουν λεπτομέρειες μάλλον είναι ένα έγκλημα μίσους ομοφοβικό σε τεράστια κλίμακα. Άρα λοιπόν αν δεν μπορούμε να επισημάνουμε ποιο είναι το πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουμε. Κύριος Ράδερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αγαπητέ συνάδελφε ε, και να ζητήσω και από τον Επίτροπο να με ακούσει. Χτες ο Πρωθυπουργό της Τουρκίας είπε πως δεν πρόκειται να αλλάξει το αντομοκρατικό της δίκαιο ούτε καν για την απελευθέρωση του καθεστώτος χορηγήσεων. Και αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τη συμφωνία μας με την Τουρκία. Τι κάνει η Κομισιόν. Έχει πλαν B για τη συμφωνία αυτή. Αν αποτύχει εάν η Τουρκία δεν σέβεται τις δεσμεύσεις της και πώς θα στηρίξετε εσείς τα κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, όπως η Βουλγαρία, στα εξωτερικά του σύνορα, σε περίπτωση που χιλιάδες πρόσφυγες φτάσουν εκεί για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Πώς θα εξασφαλίσετε περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ μυστικών υπηρεσιών έτσι ώστε να αποφύγετε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Και τέλος, ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο ασφαλής αν η Βουλγαρία μπει στο Σέγγεν. Και με τον τρόπο αυτό έχει και απόλυτη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τότε η μάχη κατά τη τρομοκρατίας θα είναι πιο αποτελεσματική. Ευχαριστούμε κυρία Πόστ. Ευχαριστώ πολλά από τα ζητήματα που ήθελα να θίξω έχουν ήδη αναφερθεί. Ήθελα παρόλα αυτά να κάνω ένα σχόλιο. Πριν από τρεις μήνες, τον Μάρτιο, ο συναδέλφός σας, ο κύριος Τηλιανίδης, μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθική υποχρέωση να δεχτεί σύρους πρόσφυγες. Και ο Πρωθυπουργός Κάμερον πρότεινε να το στέλνουμε πίσω στην Τουρκία όλους. Και η Επιτροπή ήταν κατά τη άποψη αυτή. Τελικά όμω τρει μήνε μετά αυτό ακριβώ κάνουμε. Στέλνουμε του πρόσφυγες τη Συρίας από την Ελλάδα προ την Τουρκία. Με ακριβώ αυτού του ανθρώπου που ήρθαν με τι βάρκε ω την ε, Ελλάδα. Τι ακριβώ λοιπόν συμβαίνει. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συζητάνε, ξανασυζητάνε, συζητάνε ποτέ τελικά πόσο έχουμε παρεκτραπεί, πόσο ξενοφοβικοί γινόμαστε και πόσο υποδαβλίζουμε αυτά τα συναισθήματα ξενοφοβίας σε όλη την Ευρώπη. Πώς βοηθούμε τις γείτονες χώρες, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της Τουρκία και προς τις δικές μου δικούς της πολίτες. Είναι ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε αμέσω. Πρέπει να δούμε πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δέχεται πρόσφυγε, όχι απλώ να του στέλνει πίσω. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ. Πόσοι άνθρωποι μετεγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, πόσοι στην Πορτογαλία, και ποια κράτη-μέλη δεν θέλησαν να υποδεχτούν ανθρώπους στα πλαίσια της μετεγκατάστασης. Ποια, σε ποια, ποια κράτη-μέλη σε ποια μελη μάλλον δεν μετεγκαταστάθηκε κανείς μέχρι στιγμής. Η κυρία Γκρίσμπακ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είχα δύο ερωτήσει, αλλά αυτή που αφορά τη γαλάζια κάρτα και το πεδίο εφαρμογή τη είναι ένα θέμα που το έφυξαν οι συνάδελφοι, το αφήνω απλώς στο λεπτό που μου αναλογεί να θίξω το θέμα του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το θέμα αυτό και όπως γνωρίζετε κύριε Επίτροπε προχωρούν καλά οι τριμερείς διάλογοι και Κάποιε ομάδε, μεταξύ των οποίων και οι δικοί μου, στηρίζαν την ιδέα ενό οργανισμού που να έχει ακόμη περισσότερο ευρωπαϊκή διάσταση. Θέλαμε τον πλήρη εξευρωπαϊσμό τη Frontex για να είναι πιο αποτελεσματική και να μπορεί να δράκε και αμέσω στα ζητήματα που μα αφορούν άμεσα. Ε, κύριε Επίτροπε, στηρίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άρθρο 18 και τι καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Διότι η λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα μέσω τη Επιτροπή. Δυστυχώ η δική σα θέση ω Επιτρόπου είναι της ομα... και ίδια της, ομα... της ομάδας μου και δυστυχώς θεωρήθηκαν απόψεις ε, μειονότητας. Το Συμβούλιο πάει πιο μακριά και σε περίπτωση αποτυχίας άρνησης ή αδράνειας ενός κράτου που τα αφορά ε, η διαπερατότητα ή το ευάλωτο των σύνορων του, εκεί μπορεί να επανέλθουν οι έλεγχοι στα σύνορα χωρίς ε, καμία δυσκολία. Αυτό λοιπόν πλήττει τα σύνορα Σέγγεν. Τι θα κάνετε, πώς θα προσπαθήσετε, πώς θα δράσετε για να προστατεύσετε τα σύνορα Σέγγεν. Το αναφέρετε και στην εισήγησή σας, είναι πολύ σημαντικό για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η κυρία Φλάιν. Κύριε Επίτροπε, Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα πολύ γρήγορη και με συγχωρείτε για του ε, διερμηνεί. Ξέρετε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση να αναθεωρηθεί ο κανονισμό του Δουβλίνου. Να απέχει πολύ από αυτό που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο στην έκθεση Κέγγια Μετσόλα για, την, ε, για το σεβασμό τη πρώτη αρχή αυτόματο μηχανισμού κατανόμη ευθυνών μεταξύ των κρατών Και ακόμη πιο σημαντικά ε, για την ανάληψη κεντρικού χαρακτήρα στην όλη διαδικασία. Ε, υπάρχει ένα διορθωτικό μηχανισμό, αλλά δεν είναι σαφέ πώ θα λειτουργεί, πώ θα ενεργοποιείται αυτομάτω και πώ θα κινητοποιείται Εάν θα τον κινητοποιούν τα κράτη-μέλη, θα είναι αυτόματο. Ε, είναι αφηρημένα και θεωρητικά τα κριτήρια και δεν λαμβάνει υπόψη τι παρούσε συνθήκε με ένα σύστημα ε, που ήδη καταρρέσει τα περισσότερα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλέ πτυχέ του προτινόμενου κειμένου που πρέπει να, να τι ξαναδούμε, διότι εγείρουν ανησυχίε για τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν για το νέο πλαίσιο εταιρική σχέση που προτείνεται, κανεί ε, δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζεται ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα για την Αφρική, όμω η πρόταση αυτή επικεντρώνεται στη διαχείριση των συνόρων και τη επιστροφή. Αυτή η αιρεσιμότητα πραγματικά προδίδει τις αρχές αναπτυξιακής βοήθειας που έχουμε αρχίσει να καταστρώνουμε για το μέλλον. Ε, η ανάπτυξη και η συνεργασία, η συνεργασία για αυτήν, για τις επενδύσεις, δεν γίνονται σωστά. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους Αφρικανούς, όχι απλώς να εκχωρούμε εξωτερικώς την, ε, την διαχείριση των συνόρων μας. Πραγματικά καημένη γερμηνή σήμερα, η κυρία Σουίνμπεργκ. Eh, ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Αβραμόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που μας ενημερώσατε. Και πρέπει να σας πω ότι πέρασαν 4,5 μήνες από την τελευταία φορά και νομίζω ότι δεν μας παρουσιάστηκε και πολλές καινοτομίες. Νομίζω ότι το ίμιση των ε, προσφύγων στην ε, Ευρώπη έχουν έρθει για οικονομικούς λόγους και δεν νομίζω ότι χρήζουν ασύλο. Και αυτό σύμφωνα με τον Φραντ Τίμερμανς. Λοιπόν, δεν είναι τυχοδιώκτες. Ε, για μένα είναι. Έχουν περάσει από 20 χώρες για να φτάσουν τη Βόρεια Ευρώπη. Στη Σουηδία να δείτε τι γίνεται. Έχουμε δει ανθρώπους που λένε ότι απογοητεύτηκαν γιατί θεωρούσαν ότι θα φτάσουν στη Σουηδία και θα τους δώσουν χρήμα και στέγη και φύγαν από τη Σουηδία γιατί θεωρούσαν πως δωρεάν θα λάβουν ό,τι επιθυμούν. Ε, ναι, αυτό για μένα είναι τυχόδιοκτισμό. Τώρα, για του μετανάστε οι οποίοι επιμένουν ε, και ότι θα ενσωματωθούν και τα λοιπά. Πόσο ακόμα θα τιμωρείτε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Πρόεδρε, κύριε Αβραμόπουλε, θα θέσω το θέμα της μετεγκατάστασης των προσφύγων από την ε, Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να μετεγκατασταθούν 60.400 πρόσφυγε. Με βάση τα στοιχεία που και εσείς έχετε δώσει έχει γίνει μετεγκατάσταση μόνο 1.503 ε, προσφύγων είχατε δεσμευτεί ότι θα γίνει μια προσπάθεια να έχουμε 6.000 μετεγκαταστάσεις το μήνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει σε πράξη. Διότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Το έχει διαπιστώσει και η ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε πριν λίγο καιρό στην Αθήνα. Επομένως το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η μετεγκατάσταση. Υπάρχουν ευθύνε στην ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν ευθύνε στην Κομισιόν. Υπάρχουν ευθύνε σε άλλα κράτη-μέλη. Ακούσαμε του συναδέλφου από την Πορτογαλία ότι η Πορτογαλία ζητά μετεγκαταστάσει και όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αυτή. Παρακαλώ να έχουμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Επίτροπε, οι συνάδελφοι πρόλαβαν. Τώρα να προλάβετε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω ε, εκφράζοντας το θυμασμό μου για τους διερμηνείς. Διότι όλοι ομιλούμε σαν πολυβόλα σήμερα. Κύρια Γκόμες, ε, κύριε Κοέλιο, θίξατε το θέμα. Ήμουν στην Πορτογαλία προσφάτως και να ξεκινήσω επενώντας και πραγματικά συγχαίροντας τη χώρα σας για την επίδειξη του πραγματικού νοήματος της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών. Αυτό εννοούμε όταν λέμε αλληλεγγύη. Υπάρχουν όμως τεχνικά και νομικά κολλήματα. Έχουμε προσφέρει πλήρη στήριξη στις αρχές και στην Ελλάδα και στην Ιταλία προκειμένου να ξεπεράσουν τα κολλήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, είναι απλώς θέμα ημερών για να κλείσει αυτό το εκκρεμέ ζήτημα. Κυρία Γκυγιόμ, συμφωνούμε. Είμαι απολύτω σύμφωνο. Ε, το να επενδύσουμε στην ένταξη θα κάνει την Ευρώπη μια πιο ε, ευημερούσα, ε, συνεκτική ε, και συμμετοχική κοινωνία. Για το κόστος της μη ένταξης, σαφώς θα είναι ψηλότερο από την επένδυση στις πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης. Όπως ξέρετε είναι από τις κορυφαίες μας προτεραιότητες. Τώρα τα κράτη-μέλη. για τι δράσει προστιθέμενη αξία που αναφέρατε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοιε προκλήσει. Δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο με προστιθέμενη αξία. Αυτό επιζητούμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να μάθουν το ένα από το άλλο. Δεύτερον, να μεταδίδουμε τις και να γνωστοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουμε τα κρατημέλη για να προάγουν την ένταξη και την κοινωνική συμμετοχή. Για τη γαλάζια κάρτα. επανελιμένος αναφέρθηκα σε αυτό στο παρελθόν. Είναι το καλύτερο παράδειγμα που έχουμε διότι αποφασίσαμε να αναθεωρήσουμε του σχετικού κανόνε για να προσαρμοστούμε στην σημερινή πραγματικότητα και στι πραγματικέ μα ανάγκε στην Ευρώπη. Η γαλάζια κάρτα πρώτα απ' όλα επινοήθηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχημένο τρόπο στη Γερμανία. Τώρα όμω πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκή πολιτική. Κοινή σε όλου. Η μεταρρύθμιση του συστήματος θα στηρίξει τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις και εταιρείε τους για να προσελκύουμε υψηλών προσόντων υπηκόους τρίτων χωρών από όλο τον κόσμο για τους τομείς αυτούς ε, στους οποίους αντιμετωπίζουμε έλλειψη εργαζομένων με προσόντα στα ερχόμενα χρόνια. Και Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας για την νόμιμη μετανάστευση. Ε, το ξέρετε και επιβεβαιώθηκε ενώπιον σας πριν από ένα χρόνο ότι η νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να είναι μία από τις μελλοντικέ μας πολιτικές. Ήδη έχουμε θεσπίσει, έχουμε λάβει μάλλον αποφάσεις για τους φοιτητές και τους ε, ερευνητές. Ε, μπορώ να πω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που μας ενθάρρυνε και μας παρότρινε να κάνουμε κάτι τέτοιο όσο το δυνατόν περισσότερο, ότι τα καταφέραμε. Το ίδιο και για τους εποχιακούς ε, εργαζομένους. Πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό και σε σχέση με όλα τα εργαλεία που έχουμε πριν μετανάστευση για τον κανονισμό Δουβλίνου. Δεν συμφωνώ μαζί σα. Είναι φιλόδοξη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Από την άλλη, θα συμφωνήσω ότι δεν πρέπει να την αποδυναμώσουμε την πρόταση αυτή. Όπως έχω πει, ε, είπα και στη Σεσίλια Δίκστρομ προηγουμένως, ότι ποιες είναι οι απόψεις μας σχετικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τα συζήτησα στον Καναδά με την κυβέρνηση της χώρας και ήταν σαφές το είπα ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις και δεν σκοπεύουμε να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε συμβιβασμού. Βεβαίως θα λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους αυτών των ζητημάτων. Όμως ήμουν επίσης τελείως σαφή ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας με συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα για να επιδιώξουμε αμοιβαία αναγνώριση των θεωρήσεων. Για τη Βουλγαρία και το Σέγγεν. Η θέση μας παραμένει σταθερή. Θεωρούμε ότι και η Βουλγαρία και η Ρουμανία πρέπει να γίνουν πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν. Θα γνωρίζετε ότι εξαρτάται από το Συμβούλιο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τελείως σαφής. Και όπως έχω ξαναπεί, τα εργαλεία του Σέγγεν και η σωστή τους χρήση πραγματικά μπορούν να συνεισφέρουν στην ασφάλεια. Κυρία Χέλτσερ, ε, για λόγους οικονομίας χρόνου θα μου επιτρέψετε να σας παραπέμψω στην έκθεσή μας που εγκρίθηκε μόλις προδιόρου, πριν την άφηξή μου εδώ πώς έχουν τα πράγματα για την μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση. Έχει σαφείς απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέσατε. Όντως, είναι κοινή μας ευθύνη το πώς θα προχωρήσουμε προς το μέλλον και το είπατε και προηγουμένως σε ό,τι αφορά τους αριθμούς και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη. Συμφωνείτε, είπατε, με τον κύριο Τίμερμαν. Όμω ο κύριο Τίμερμαν συμφωνεί μαζί μου. Άρα, κατ' επέκταση και κατ' επαγωγή, συμφωνείτε και μαζί μου. Κυρία Γκρίσπεκ, δεν χρειάζεται να πρασπιστώ τη θέση τη Επιτροπή. Το γνωρίζετε. Η πρότασή μα, όπω πολύ σωστά είπατε, είναι αυτή. Λυπούμε που η πλειοψηφία της Επιτροπής αυτής δεν στήριξε την πρόταση της Επιτροπής. Κατανοώ ότι οι τριμερείς διάλογοι δεν έχουν φτάσει στην εξέταση του άρθρου 18 και πραγματικά αναμένω με ανυπομονησία να φτάσουν ως εκεί. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω λίγο ελληνικά, γιατί μου έθεσε ένα ερώτημα και ο κύριο Μαριά. Πού πήγε. Α, ωραία. So, let me do it in Greek. Στα ελληνικά, παρακαλώ. Για λόγους ευγένεια. Θέλω να ε, παραπέμψω τον κύριο Μαριά, όπως ανέφερα πρωτήτερα, στο report που όπως είπα πριν μόλις υιοθέτησε. Welcome. Καλώς ήρθατε κύριε I Στο report που μόλις υιοθέτησε η Επιτροπή για το State of Play στην μετεγκατάσταση και ε, ήθελα να σας πω ότι μέσω αυτού στείλαμε ξεκάθαρα συγκεκριμένα μηνύματα προς όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους. Σας είπα στην αρχή ότι πλησιάζει η ώρα πλέον να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σύντομα, εάν δεν υπάρξει πρόοδος μέσα στις προσεχείς ημέρες, θα αναγκαστώ πλέον να πω ονόματα και διευθύνσεις. I intend to name and shame. Και συμφωνώ με τη γενική παρατήρηση που έκαναν όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς, ότι είναι η στιγμή που κρίνεται στην πράξη η δυνατότητα και η θέληση να αποδείξουμε όλοι ότι το εννοούμε όταν μιλάμε για υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Και κάτι τελευταίο. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε δουλέψει πολύ εμείς και λέω εμείς, η Λίμπε Κομίτη, η Κομισιόν και εγώ προσωπικά μαζί σας. Και δεν θέλω να σας κολακέψω, αλλά το έλεγα πρωτήτερα ότι από την αρχή έμαθα πολλά κατάλαβα περισσότερα και ενθαρρύνθηκα από εσά για να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Δεν θα συμφωνήσω όμω με τι παρατηρήσει ότι δεν έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη πριν από 1,5 χρόνο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προβλημάτων. Και αναφέρομαι και στην ασφάλεια και βεβαίω κυρίω στη μετανάστευση. Τώρα υπάρχει πλαίσιο, υπάρχουν αρχέ Υπάρχει στρατηγική, το κυριότερο όμως από την πλευρά μας, υπάρχει η πολιτική βούληση να συμβάλλουμε μαζί με όλους τους παράγοντες, τόσο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω, διότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, παγκόσμιο το θέμα και το οποίο θα μας συνοδεύει και εμάς και τα επόμενα κοινοβούλια και τις επόμενες επιτροπές, γιατί φοβούμε ότι θα κρατήσει για πολλά χρόνια αυτή η δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Και η Ευρώπη ετοιμάζεται. Τα όσα σήμερα είπαμε και έχουμε πει κατά καιρού, το αποδεικνύω και σας ευχαριστώ πολύ, διότι είναι η Επιτροπή που στην ουσία είναι ο κατεξοχήν συνομιλητής τη Επιτροπή και η οποία μας έχει βοηθήσει και το αναγνωρίζουμε δημόσια και σας μόνο για αυτό. Thank you very much for your attention. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Είδατε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για συζητήσεις μαζί σας. Ευχαριστούμε συνάδελφε για τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας. Ε, είχαμε πίεση χρόνου και τώρα να αφήσουμε τον Επίτροπο να φύγει στην ώρα του. Now, uh, we will as the colleague ah, Mr. is present. Α, ο κύριος Μπόρνη είναι εδώ. Οπότε να ξεκινήσουμε και μαζί σας. So the next point on our agenda... Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. είναι το ζήτημα των νέων ψυχότροπων ουσιών. Έχουμε τον κύριο Μπόρνη και μόλις έρθει η κυρία Βάριο, η οποία δεν είναι εδώ σήμερα όμως. Έχουμε τον κύριο Μπόρνη, τον εισηγητή της δέσμης μέτρων για, τα, για τις νέες ψυχότροπες ουσίες, ο οποίος θέλει να ενημερώσει σήμερα την Επιτροπή μας για την επίκαιρη κατάσταση. Είμαι σίγουρη πως πολύ θέλετε να φύγετε, αλλά παρακαλώ φύγετε ήσυχα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Μπόρνη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την επικύρη κατάσταση μετά την απόφαση με τον σκιώδη συγκητή κύριε Μπόνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εκ μέρους της Τερέσα Χιμένες και από μένα θα ήθελα να σας ενημερώσω για την επικύρη κατάσταση της εργασίας επί της νέας δεσμής μέτρων για νέες ψυχότροπες ουσίες. Η Τερέσα είναι η εισηγητρία με αντικείμενο την θέσπιση ελάχιστων διατάξεων Σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, μια στιγμή, μια στιγμή, παρακαλώ, διακόπτη ή προεδρεύουσα. Αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ, να αποχωρήσουν τώρα, επειδή έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Σας ενημερώνω πως παρουσιάζω την επικυρή κατάσταση των εργασιών σχετικά με την έδεσμη μέτρων για ψυχότροπες ουσίες εκ μέρου μου και τις τέρες αχημένες. Η Χιμέσα είναι η εισηγήτρια της οδηγίας και θέτει ελάχιστε διατάξεις σχετικά με την υπόσταση έγκληματων και ποινών που ισχύουν στον τομέα της παράπονης διακίνησης ναρκωτικών. Όσον αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών, και εγώ είμαι ησυχητής για τον κανονισμό για νέες ψυχοτροπές ουσίες. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις πληροφορίες αυτές, όχι μόνο εκ μέρους της Τερέσα, αλλά εκ μέρους όλων των σκιωδών. Εμείς όλοι οι σκιώδεις συναντήσαμε την Ολλανδική Προεδρία και την Κομισιόν τον Απρίλιο του 2006 και ενημερωθήκαμε πως το Συμβούλιο προτίθεται να εγκρίνει μια κοινή θέση, την κοινή θέση με μια μικρή απόκληση. Θα ήθελα να σας θυμίσω πως εγκρίναμε την τοποθέτησή μας την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο και έκτοτε περιμένουμε το, την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Η διαδικασία ήταν μακρά μέχρι να βρεθεί μια λύση στο Συμβούλιο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που αυτό απετεύχθη. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή μας παρουσίασαν την προσέγγιση αυτή και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λαμβάνοντας υπόψη την επίγουσα ανάγκη νομοθεσίας στον τομέα αυτό και των δυσκολίων που επέφερε η προηγούμενη προσέγγιση καθώς δεν μπορούσε να, να βρεθεί μια κοινή λύση κατά τη διάρκεια του τριμερού λόγου, οι σκιώδεις πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν αυτή τη νέα προσέγγιση για, το, για τη δέσμη μέτρων και να συνεργαστούν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να επιτύχουν μια συμφωνία η οποία θα μπορεί να εγκριθεί το γρηγότερο δυνατόν. Η νέα προσέγγιση θα περιλαμβάνει τη διεύρυνση της οδηγίας βάσει του άρθρου 83 της συνθήκης με τις διατάξεις της ανταλλαγής πληροφοριών, την εισαγωγή δύο κατηγοριών κινδύνου ως προς την εκάστοτε ουσία, τη λήψη περαιτέρω δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε προηγούμενες λύσεις είχαμε τρία επίπεδα κινδύνου εάν η ουσία αξιολογηθεί ως επικίνδυνη, η ουσία αυτή θα υποκείται σε διαρκή μέτρα ελέγχου με τη μορφή μιας πανενοσιακής υποχρέωσης να κηρυχθεί η ουσία παράνομη σε εθνικό επίπεδο. Οι διατάξεις του συστήματος πρώιμης προειδοποίησης και ανάλυσης κινδύνου και αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στον προτινόμενο κανονισμό θα συμπεριλάβουν περαιτέρω μέτρα όσον αφορά τον κανονισμό περί MCDA και η αναθεώρηση του κανονισμού αυτό θα περιοριστεί μόνο στο στοιχείο αυτό και θα αποτελέσει τμήμα της όλης δεσμής μέτρων. Αυτό είναι μια δυνατότητα για όλους μας να συνεχίσουμε την εργασία μας, να έχουμε ταχύτερα αποτελέσματα επειδή τώρα έχουμε μια κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και επιτύχαμε πρώτον το σύστημα πρώιμης προειδοποίησης και ένα νέο μοντέλο απαγόρευσης της εμπορίας και της χρήσης τέτοιων ουσιών σε όλη την Ευρώπη με έναν κάπως διαφορετικό τρόπο από ότι αυτός προτάθηκε στην προηγούμενη λύση. Λοιπόν, οι στόχοι είναι πολύ κοντά, αλλά πρέπει να αλλάξουμε την εργασία μας και είμαστε ανοιχτοί, εγώ, η Τερέσα φυσικά και οι σκιώδεις εισηγητές, μετά από τις ε, συζητήσεις μας για να προχωρήσουμε. Ο κύριος Μπόνη, κύριε Μπόνη, συγγνώμη. Δεν βλέπω κάποιον σκιώδη εδώ. Θα ρωτήσω του συναδέλφου αν θέλουν να παρεύουν. Αν όχι, θα ζητήσω από την κυρία Σίπαλα, εκ μέρου τη Επιτροπή, αν θέλει να επέμβει, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Επίση, επειδή κατανοώ πω ε, και η Προεδρία βρίσκεται εδώ και θέλει να πει κάτι, θα ήθελα να ευχαριστήσω του σκιώδε και του εισηγητέ για την αποφασή του. Προσδοκούμε να συνεργαστούμε με περισσότερη ταχύτητα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για τη νέα προσέγγιση αυτή, την οποία υποστηρίζει η Επιτροπή υπό ορισμένους όρους. Γι' αυτό και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να υλοποιήσουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από τη Συμφωνία. Και έτσι ώστε η Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μπορέσει να επιτυχεί πρόοδο. Οπότε δίνω τον λόγο στην Ολλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπόνη. Το, στο Συμβούλιο αποφασίστηκε μια προσέγγιση που μας παρουσίασε ο κύριος Μπόνη και είμαστε ευχαριστημένοι που το Κοινοβούλιο θέλει να εργαστεί με βάση αυτό. Η Προεδρία εργάστηκε για να προχωρήσει η εργασία όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν έχουμε προς το παρόν μια γενική προσέγγιση, αλλά τη σκιαγράφηση, η οποία θα αποτελέσει την βάση για την εργασία στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπόνη. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη συνεργασία της και ιδίως την Ολλανδική Προεδρία. Επειδή συνεργαστήκαμε με διάφορες προεδρίες τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά από ό,τι αποδειχθήκε η Ολλανδική Προεδρία είναι η πιο αποτελεσματική για την επίτευξη αυτή τη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω η συμφωνία να είναι επιτυχής. Και τώρα θα επιστρέψουμε, ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχω το σημείο 12. Παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Το σχέδιο δράσης αυτό παρέχει ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής και μέτρα στα κράτη-μέλη για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών οι δράσεις που προτείνονται στο σχέδιο της Επιτροπής βρίσκονται σε βασικούς τομείς όπως είναι η πρώιμη ένταξη, ιδίως για ανθρώπους που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, την πρόσβαση στην, στην εκπαίδευση, σε βασικές υπηρεσίες και την κοινωνική ένταξη. Το σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση του υφιστάμενου πλαισίου για την ένταξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ένταξης με την οποία σχετίζεται η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια σε όποιον θέλει να παρέμβει εκ μέρους της Επιτροπής, ο κ. Σάβαρη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω το σχέδιο δράση αυτό σχετικά με την ένταξη υπηκών των χωρών. Λίγε λέξει πρώτα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο τη Επιτροπή, γιατί όλοι γνωρίζουμε και το γνωρίζετε κι εσεί πολύ καλά ότι στον τομέα αυτό τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πολλέ προκλήσει στον τομέα τη ένταξη λόγω των ε, εισρώων επικόντρων χωρών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρήσαμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να επενδύσουμε στην ένταξη και όπω είπε προηγουμένω και ο Επίτροπο ε, στην παρέμβασή του, το κόστο τη μη ένταξη ε, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το να επενδύσουμε τώρα σε πολιτικέ ε, σωστή ένταξη. Η ένταξη είναι έτσι κι για μια συνεκτική και συμμετοχική κοινωνία και είναι κοινή ευθύνη όλων των ε, φορέων κρατών μελών που έχουν την ύψιστη αρμοδιότητα σε αυτόν τον τομέα, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και Αυτή η φιλοδοξία είναι και κατανοητή. Για πρώτη φορά καταφέραμε να έχουμε με αυτό το πρόγραμμα την ένταξη ως ένα πρωταρχικό ζήτημα καθότι πολλές πολιτικές μπορούν να συνεισφέρουν στην ένταξη. Η απασχόληση, τα βλέπουμε με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και στο πρόγραμμα δράσης, υπάρχουν πολλές αναφορές στο νέο θεματολόγιο για, τα, για τις δεξιότητες, Επίσης, για την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, στις περιφερειακές πολιτικές που τις αφορά η διάσταση της ένταξης επίσης. Είναι λοιπόν φιλόδοξη, ε, συνολική αλλά και συγκεκριμένη η πρότασή μας, διότι η ανακοίνωση αυτή με το πρόγραμμα δράσης ε, δεν είναι τελείως θεωρητική μόνον αλλά έχουμε συμπεριλάβει στο παράδειγμα 15 και συγκεκριμένε δράσει, οι οποίε είναι εργαλεία τα οποία προτείνονται στα κράτη-μέλη για να τα στηρίξουμε στι δράσει ένταξη. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε χρηματοδότηση, οι οποίε θα προταθούν στα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών και τι οργανώσει τη, που ενεργοποιούνται στον τομέα τη ένταξη τα ερχόμενα χρόνια και θα δείτε ότι σκοπεύουμε να ενισχύσουμε το δίκτυο των εθνικών υπευθύνων για την ένταξη. Θα προσπαθήσουμε να το μετατρέψουμε σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την ένταξη, για το οποίο βεβαίως θα ενημερώνονται διαρκώς και η Επιτροπή Λίμπε και η Γραμματεία της, όπως και τώρα συμβαίνει. Και τώρα ας δούμε το περιεχόμενο του προγράμματος. Έχουμε πέντε περιοχές στόχους. Πρώτη, η τα μέτρα πρώτης άφηξης, πρώτης αναχώρησης, μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν ήδη σε τρίτες χώρες προέλευσης για να προετοιμαστεί η έλευση των ε, μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με μαθήματα ενδεχομένω, μέτρα τέτοιου τύπου, επί τα μέτρα για την ε, ενημέρωση περί της κοινωνίας στην οποία θα φτάσει ο μετανάστης. Αυτά βεβαίως ε, κυρίως μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση της μετακατάστασης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη προτεραιότητα, η εκπαίδευση. Συνεργαστήκαμε για αυτά με, την Γενική Διεύθυνση, με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Βεβαίως, εδώ αυτό θα έχει τεράστια επιρροή στη χάραξη πολιτικής και έχουμε πολλά σχετικά εργαλεία για την ένταξη, ιδίω έλεγχο των γλωσσικών ικανοτήτων των αφιθέντων μεταναστών online, της ε, πλήρως ε, ε, συνεκτικής εκπαίδευσης για όλους τους μετανάστες με τη συμπερίληψη των παιδιών των μεταναστών στην προσχολική εκπαίδευση ήδη και έχουμε μία ως δυνατόν πιο σφαιρική προσέγγιση, ιδίως σε αυτό το τομέα. Τρίτος τομέας προτεραιότητας ένταξη στον τομέα απασχόλησης και εργασίας και επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις με το θεματολόγιο για τις δεξιότητες που πρόσφατα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προωθηθεί ταχύ διαδικασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε οι μετανάστες να έχουν πρόσβαση στην αγορά πολύ γρήγορα και να ε, ε, αυτή τη στιγμή εγκριθεί το καθεστώ του. Επίση, η αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων, που μέχρι τώρα είναι ένα πρόσκομα για την πρόσβαση στην αγορά και επίσης οι ασκήσεις και οι μαθητείες των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθηθούν με όλες τις βελτιστές πρακτικές και τις τεχνικές που αναλογούν και πρέπει να παρατηρηθούν τα κάτω να αναπτύξουν. Άλλο σημαντικό τομέα είναι πρόσβαση στι βασικέ υπηρεσίε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τόσε αρμοδιότητε, διότι αυτά επιλύονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στον τομέα αυτό. Αλλά προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε την πρόσβαση στι βασικέ υπηρεσίε για του υπηκόρου τρίτων χωρών. Όλο ιδιαίτερο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει ήδη προσφέρει πολλά δάνεια για να βελτιώσει τι δυνατότητε υποδοχή κρατών μελών στον τομέα αυτό. Επίση, στον τομέα τη υγεία, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένη μαθητεία για τους επαγγελματίες του χώρου, ώστε να καλύψουμε τις ειδικέ ανάγκες των και τρίτων χωρών στον τομέα αυτό. Τελευταίο και εξίσου σοβαρό, επικεντρωθήκαμε στο πρόγραμμα δράση και στην ενεργό συμμετοχή τη κοινωνική συμμετοχή και ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών, προκειμένου να προωθηθούν οι ευρωπαϊκέ αξίε, ο διαπολιτιστικό διάλογο και η γνωστοποίηση των ευρωπαϊκών βασικών αξιών. Οι αθλητικέ δραστηριότητε, οι πολιτιστικέ δραστηριότητε, οι εκδηλώσει είναι πολύ σημαντικέ για του μετανάστε και επίση στηρίζουμε την προώθηση δράσεων για την καταπολέμηση τη διακριτική μεταχείριση και την ξενοφοβία καθώ και το ρατσισμό. Υπάρχουν και δύο οριζόντια σημεία στα οποία ήθελα να επιμείνω στο πρόγραμμα δράση. Η χρηματοδότηση, που ξέρετε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο, εφόσον δεν έχουμε δυνατότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναλάβουμε νομοθετική δράση στον τομέα τη μετανάστευση απευθεία. Μπορούμε όμω να στηρίξουμε αυτέ τι δράσει με τη χρηματοδότηση. Έχουμε συγκεκριμένο κεφάλαιο γι' αυτό, ε, με τίτλο Τα κονδύλια. Και ε, αυτό για να στηρίξουμε την μετανάστευση επικόντρων χωρών και τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Υπάρχει επίση ένα τμήμα για τον καλύτερο συντονισμό, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων και των θεσμικών οργάνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα δράση. Νομίζω αυτά ήταν τα βασικά σημεία που ήθελα να υπογραμμίσω για αυτό το πρόγραμμα δράση. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμεί ευχαριστούμε. Η κυρία Λαουρίστα έχει Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και νομίζω ότι τέτοιου είδους σχέδια δράσης είναι πολύ σημαντικά γιατί έχουμε συζητήσει θέματα ενσωμάτωσης και είναι καλό να έχουμε και κάποια συγκεκριμένα βήματα μπροστά μας. Έχω λοιπόν μια ερώτηση να σας κάνω. Ξέρετε καθόλου πού μπορώ να βρω αυτή την το προφίλ των όσων εισέρχονται, δηλαδή ε, τι παιδεία έχουν, ε, τι προσόντα έχουν κτλ. Γιατί ένα τέτοιου είδους προφίλ μας βοηθά ε, στο να βρούμε και τα μέσα για να καλύψουμε τις ανάγκες του. Να δούμε αν για παράδειγμα κάποιοι είναι δάσκαλοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα σημεία που λείπει από την συγκεκριμένη αυτή παρουσίαση. Χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες. Η κυρία Ζήπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως το ζήτημα της ένταξης είναι κεντρική σημασίας. Ωστόσο, επίσης ένα θέμα στο οποίο τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε προβλήματα αρχής. Αναφέρομαι παραδείγματο χάρη στην ένταξη ανθρώπων με αναπηρίες, στην ένταξη των Ρωμά και πολλών άλλων ομάδων, τότε έχουμε ήδη ένα εσωτερικό πρόβλημα ένταξης σήμερα το σκεπτόμασταν, σκεπτόμασταν πως επρόκειτο για έναν τομέα καθηκόντων που ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και έναν εντονότερο εξευρωπαϊσμό στον τομέα αυτό. Όσον αφορά τους ανθρώπους από τρίτους χώρες, έχουμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία όσον αφορά την ένταξή τους, όσον αφορά παραδείγματος χάρη την εκμάθηση της γλώσσας, αλλά επίσης σημαντικές γνώσεις για την καθημερινότητα. Οπότε προκύπτει το ζήτημα του πόση προσαρμογή χρειάζεται, ποια προσόντα χρειάζονται, ποιε δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία άρχισαν στα, κράτη, στα πλαίσια της καταχώρησης των προσφύγων κατά την είσοδό τους να καταχωρούν επίσης τέτοια στοιχεία έτσι ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν χρειαστεί. Οπότε υπήρξαν οι σκέψεις κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει στα πλαίσια της επανεγκατάστασης. Θα ήθελα όμως καταρχάς στο θέμα της ένταξης να μην παραμείνω στους πρόσφυγες. Έχουμε επίσης προτάσεις για τη διεύρυνση της νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, η οποία δεν περιορίζεται σε ακαδημαϊκά επαγγέλματα, επειδή στα ευρωπαϊκά κράτη μας έχουμε ζήτηση σε πολλούς διαφορετικούς τομείς αλλά ακόμα και εκεί πρέπει να αποσαφινιστεί ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια αναγνώριση μπορεί να χορηγηθεί και εκεί θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι σε τρίτες χώρες για τη δυνατότητα εργασίας εδώ σε εμά, ποια είναι η συνεργασία με τα κράτη προέλευσης, τι μπορεί να γίνει εκ των προτέρων, ιδίως κατά την εκμάθηση της γλώσσας, και πού βρίσκεται το ευρωπαϊκό καθήκον. Υπήρξαν ήδη συνομιλίες με τα κράτη-μέλη. Σε ποιο έδρος και σε ποιους τομείς με κράτη-μέλη τα οποία διατίθεται να προβούν σε συγκεκριμένα μέρη για το ζήτημα της ένταξης. Η κυρία Σπινέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή <clears throat> για τη σχέση μεταξύ ένταξης, ε, συστήματος υγείας και νομοθεσίας περί αγοράς εργασίας. Το ερωτώ, διότι μεγάλο μέρος των φόβων που υπάρχουν στα κάτι μέλη και ιδίως στα λαϊκά στρώματα, ο φόβος για τους μετανάστες, είναι φόβος ότι θα χάσουν δικά τους δικαιώματα οι άνθρωποι σε σχέση με το κράτος πρόνοιας. Και ότι υπάρχει εδώ ένας ε, ανταγωνισμός που θα υποβαθμίσει τις συνθήκες στην αγορά εργασίας με την αύξηση του αριθμού μεταναστών. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά αυτός είναι ο φόβος που διακατέχει τους ανθρώπους. Η ερώτηση λοιπόν που θέλω να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξή. Δεν είναι αρμοδιότητα μόνο των κρατών μελών η ε, ονομοθεσία περιεργασία και το εργατικό δίκαιο. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας και αυτή η κούρσα προς τις επισφαλείς συνθήκες του κόσμου της εργασίας είναι κάτι που ζητάται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από τα κράτη-μέλη. Το ζητάνε στα ευρωπαϊκά εξάμεινα, το ζητάνε στις επιστολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τα κράτη, που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες μεταξύ των οποίων και το δικό μου, η Ιταλία. Αυτό που τους ζητούν είναι μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, που εν γέννη πηγαίνει προς τις επισφαλείς συνθήκες, την επισφαλή εργασία. Γι' αυτό και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζοντας ότι η απάντηση δεν θα είναι απλώς αυτά είναι αποφάσεις των κατών διότι δεν ισχύει πλέον. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και με συγχωρείτε που έφτασα ε, με καθυστέρηση και που δεν κατάφερα να ακούσω και τα εισαγωγικά σας σχόλια. Είμαι πάρα πολύ δεμένη με το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία θα πρέπει να ξαναδούμε για το θέμα αυτό. Ζητώ στατιστικά στοιχεία για να μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί στη Γαλλία διαβάζουμε πολλά άρθρα για το τι συμβαίνει στη Γερμανία και πολλά είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Δηλαδή, γενικά όλες οι μελέτες εξηγούν πως οι μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και πιο εκπαιδευμένοι, έχουν δηλαδή όλο και περισσότερη παιδεία και βέβαια υποαπασχολούνται σε σχέση με την εργασία που θα μπορούσαν να εκτελέσουν. Και έχουμε μία μελέτη στην Γαλλία τελείως διαφορετική από αυτή για τους σύρους που φτάνουν. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν και είναι πολύ σημαντικό για να είναι καθαρή η ματιά μας στο θέμα. δεν μου αρέσει ε, να πιο ε, καζολιστικά επιχειρήματα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μου πείτε τι γίνεται και πολλές μελέτες αποδεικνύουν πως πολλά κρατημέλη χρειάζονται μετανάστες. Θα ήθελα λοιπόν να μου τα πείτε πιο ξεκάθαρα και να δούμε πώς μπορούμε να προκρίνουμε την ενσωμάτωση, να την ευνοήσουμε υπό τις σωστές συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες και κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις οι οποίες είναι αναντίστοιχες με τα προσόντα τους και δεν είναι στην ε, κατάσταση ε, που θα έπρεπε να είναι, όπως είπε η Μπάρμπαρα Σπινέλη, θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοίχηση μεταξύ προσόντων και εργασίας και βλέπουμε ότι πάρα πολλοί με πολλά πτυχία εργάζονται στον κλάδο των υπηρεσιών υπό συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά δραματικές. Θα ήθελα λοιπόν, εάν θέλουμε να βγούμε από τα, από στερεότυπα και να ευνοήσουμε ε, την ενσωμάτωση όχι μόνο των προσφύγων αλλά και των μεταναστών, πως θα πρέπει να έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο σε σχέση με τα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα και όχι να αντιμετωπίζουμε φαντάσματα και φόβους. Ευχαριστώ κυρία Βεζία. Ε, η κυρία Σαμερή έχει το λόγο και πάλι. Ο κύριος Σαβαρή, ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για την πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά την διάστρωση του πληθυσμού που έρχεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που τέλος πάντων ήρθε το 2014 και 2015 κυρίως, υπάρχουν μελέτες που εκπονήθηκαν κυρίως στην Γερμανία και τη Σουηδία. Ε, αυτές οι δύο χώρες δέχτηκαν το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών, ε, του, τον άσυλο μάλλον, και όπως σωστά επιδείχθη από την κυρία Γκυγιόμ, αυτό δείχνει ότι πράγματι όποια και να είναι τα προσόντα των ανθρώπων αυτών, εάν το συγκρίνουμε με προηγούμενε περιόδου μετανάστευση. σίγουρα οι αριθμοί του είναι μεγαλύτεροι. Έχουμε κάποιες μελέτες που εκπονήθηκαν, ε, μπορώ να σας αποστείλω τις σχετικές παραπομπές μέσω της γραμματείας σας, εάν ενδιαφέρεστε, και να σας δώσουν ακριβώς ε, τις παραπομπές. Τώρα, το θέμα της ένταξης ολόκληρων ομάδων, όπως είπε η κυρία Ζίπελ, Ρωμά ή ανθρώπων με δικές ανάγκες, όντως το πρόγραμμα δράσης υπάρχει ένα ειδικό εδάφιο για το θέμα αυτό, που δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ένταξη των επικών τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των ευάλωτων ή ευπαθών ομάδων ή μειονοτήτων. Δεν σημαίνει ότι επειδή θέλουμε να επικεντρωθούμε στους επικόστοι των χωρών θα παραγωνίσουμε άλλες ομάδες. Αυτό δηλώνεται σαφώς στο πρόγραμμα δράσης. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εργασίας και της μετανάστευσης, ναι, περισσότερα προσόντα και δεξιότητε τα χρειαζόμαστε. Το ξέρουμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απλώ θα παραθέσω το στοιχείο τη ανακοίνωση τη 6 Απριλίου, ανακοίνωση 6 Απριλίου πριν δημοσιευτεί η επισήμωση ανακοίνωση για το άσυλο. Υπήρχε εκεί ένα σχόλιο και για τη μετανάστευση και υπάρχουν αρκετέ σημαντικέ πληροφορίε για το θέμα τη νόμιμη μετανάστευση, για το πώ τη βλέπουμε και τι σκοπεύει να κάνει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προσεχή μήνε. Ναι, εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε γυράσκοντα πληθυσμό και ήδη έχουμε κάποια προβλήματα σε συγκεκριμένου τομεί. Θα έχουμε μεγαλύτερα τα ερχόμενα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να προετοιμαστούμε και να θεσπίσουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα νόμιμης μετανάστευσης. Διότι θα αντιμετωπίσουμε έλλειψη επαγγελματικών προσόντων ακόμα και αν λάβουμε υπόψη την ηλικία των Ευρωπαίων εργαζομένων, να αυξήσουμε τα προσόντα των Ευρωπαίων πολιτών ή αυτών που ήδη κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι θα καλύψουμε το χάσμα που θα έχουμε σε 10-20 χρόνια. Και κάτι επί το οποίο θα εργαστούμε ε, όλος ιδιαιτέρως, ενισχύοντας τις οδηγίες για την νόμιμη μετανάστευση, με αυτόν τον έλεγχο υγείας, τον οποίο θα ακούσει το check-up, το fitness check, αυτό που αναφέρεται για να δούμε κατά πόσον λειτουργεί σωστά το κεκτημένο για τη μετανάστευση, που υπάρχουν κενά ελλείψεις και να ε, προλάβουμε να καλύψουμε ανάγκες ως προς τη μετανάστευση. Επίσης, θα διεξαχθεί μελέτη, αναφέρθηκε και αυτό στην ανακοίνωση της 6 Απριλίου, για να ε, δούμε κατά πόσον μπορούμε να προβλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σύστημα το οποίο να συνδυαστεί με το ανάλογο σύστημα του Καναδά και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τον αριθμό υπηκών τρίτων χωρών που έρχονται προ την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ανάγκες της αγορά εργασίας, ώστε να καλυφθεί και η διάσταση τη απασχόληση. Επίση, για το πώς συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο τη ε, εξακολούθηση τη Συνόδου τη Λαβαλέτα. Προσπαθούμε στον τομέα της νόμιμης, ε, της νόμιμης μετανάστευσης από τρίτες χώρες να πάρουμε πρωτοβουλίες και να αποσπάσουμε δεσμεύσεις από τις τρίτες χώρες. Δεν μπορώ όμως να πω πολλά σχετικά, γιατί η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, μάλλον μόλις ξεκίνησε. Επίσης, υπάρχει προφανώς ο φόβος του να χάσει κανείς τα δικαιώματα και να υποβαθμιστεί για τους Ευρωπαίους πολίτες και ε, αυτό εννοείται ότι το έχουμε θίξει στο θεματολόγιο, στην ανακοίνωση μάλλον, αλλά το θεματολόγιο ακριβώς για τις δεξιότητες προβλέπει την κάλυψη των δεξιότητων των Ευρωπαίων πολιτών και την ε, βελτίωσή τους για να μπορέσουν να διεκδικούν αποτελεσματικότερα μια θέση εργασίας. Και αυτό που ενδιαφέρει του υπηκόου των χωρών σε αυτό το θεματολόγιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή κοιτάζει την έγκριση των επαγγελματικών προσόντων που θα μπορούσε να αφορά το σύστημα που δημιουργείται και του υπηκόου των χωρών που έρχονται στην Ευρώπη. Μπορεί να αναγνωριστεί δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επαγγελματική του πείρα. Αυτό είναι κάτι που θα το καλύψει το θεματολόγιο για τι δεξιότητε, τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτά νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις αυτές. Συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε. Το επόμενο σημείο που έχουμε να δούμε έχει αναβληθεί. Ήταν ε, η ερώτηση Κοράου και έχουμε το τελευταίο σημείο στη σημερινή ημερήσια διάταξη που είναι μια παρουσίαση μία μελέτης την οποία ζήτησε ε, το τμήμα ΓΑΜΑ ε, Συγγραφής Πολιτικής για να, για να δούμε ποια είναι η δυνατότητα διεύρυνσης νέων οδών για την νομοθεσία σχετικά με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μαζί μας εδώ τον καθηγητή Ιβάν Μαρτίν από το Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ρόμπερτ Σούμαν, ε, από το Κέντρο Προηγουμένων ε, Μελετών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου από τη Φλωρεντία. Του δίνω λοιπόν το λόγο. Κύριε Μαρτίν, μπορείτε να μας παρουσιάσετε αυτή την ε, μελέτη και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να συζητήσουμε. Έχετε χρόνο. Γύρω στα 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τις υπηρεσίες σας που μας καλύψατε ε, ε, και που μας καλέσατε σημερινή συνεδρίαση για να παρουσιάσουμε εδώ τους νέους μηχανισμούς και τις δυνατότητες που υπάρχουν για νομοθεσία, για μια νέα εργατική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βασίζεται και σε μετανάστες. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που δεν λειτουργεί. Έχουμε μια μελέτη που τελείωσε το φθινόπωρο του 2015 ε, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πολύ επίκαιρη αυτή η μελέτη και πολύ σχετική και κυρίως σήμερα έχοντας ακούσει τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο ο οποίος παρουσίασε εδώ το νέο πακέτο για την νόμιμη μετανάστευση και άλλα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τα όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Ιουνίου έχω να σας πω πως στη μελέτη τη δική μας έχουμε εδώ τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρουσίασή μου θα δείτε τα έξι κεφάλαια ερευνά και ερωτήσεων που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε eh, και τηλεγραφικά θα απαντήσω σε κάθε ένα από τα έξι κεφάλαια. Γιατί είναι απαραίτητη μια πολιτική μεταναστευτική και εργασιακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκή. Γιατί, Γιατί έχουμε μια ενιαία αγορά εργασίας, παρόλο που ακόμα υπάρχουν πάρα, πολλά, ε, πάρα ε, πάρα πολλά στοιχεία που προέρχονται από το γεγονό ότι είχαμε 28 αγορέ εργασία. Έχουμε λοιπόν αυτά τα κληροδοτήματα που όμως παρόλα αυτά μας έχουν οδηγήσει σε μία ενιαία αγορά εργασία και έχουμε και δημόσια Ινστιτούτα και ε, πανεπιστήμια που συνέχεια παρουσιάζουν μελέτε για το γεγονό πω σπανίζουν τα χέρια ε, το εργατικό δυναμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε μάλιστα και τι 10 σελίδε τη μελέτη μα, που λένε το εξή πω όντω χρειάζεται ε, εργατικό δυναμικό και σήμερα και στο μέλλον και θέλουμε και υψηλών προσόντων και ε, ανθρώπου χωρί πολλά επαγγελματικά προσόντα ανειδίκευτους εργάτες δηλαδή. Ας δούμε λοιπόν τα διάφορα εργαλεία και τις διάφορες φάσεις από το νομικό πλαίσιο για την εργασιακή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως εδώ τα πράγματα είναι κατακαιρματισμένα και υπάρχει ένα missing link, ε, ένα κομμάτι της αλυσίδας που λείπει στην πολιτική αυτή, που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ε, υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι νόμιμα διανέμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Επίσης το τέταρτο στο οποίο θα σταθώ είναι το τέταρτο κεφάλαιο που είναι οι επιπτώσεις τη μεταναστευτική εργασία ή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά εργασία και η ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασία. Και εδώ το συμπέρασμα είναι που είναι πολύ χαμηλή η επίπτωση, σχεδόν ε, γύρω στο μηδέν, για του λόγου που προανέφερα. Κατακαιρματισμένη πολιτική που δεν αφήνει περιθώριο λιγμών στα κράτη-μέλη. Πέμπτο, Θέλαμε να δώσουμε μία απόκριση στην ερώτηση το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση που ε, δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2015 αποκρίνεται ή όχι στις ανάγκες που έχουμε να νομοθετήσουμε για τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάντηση είναι πως δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας και τέλος κάνουμε και μία γρήγορη ανάλυση τεχνικών ζητημάτων. Κοιτάξαμε 12 δυνατούς μηχανισμούς, πιθανούς μηχανισμούς ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προτείνουμε τι θα μπορούσε να κάνει. Να πω στα γρήγορα πως ε, τα συμπεράσματα που είναι σχετικά για τη σημερινή κατάσταση από την ε, έκθεση αυτή είναι το κατά πόσο είναι επίκαιρη η έκθεση αυτή. Να σας πω πως η αναθεώρηση της οδηγίας για τη γαλάζια κάρτα θα δείτε αριστερά στη στήλη πως έχετε εκεί τις τέσσερις μεγάλες προτάσεις που υποβάλλουμε για την μεταρρύθμιση της οδηγίας αυτής την αναθεώρησή της, το προτείνουμε ήδη στην ε, έκθεση και δεξιά θα δείτε ποιες είναι οι αλλαγές που εισάγονται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επαναλαμβάνω τις 7 Ιουνίου τρέχοντος. Προτείναμε λοιπόν εμεί μια μοναδική γαλάζια κάρτα που θα έδινε πρόσβαση σε όλη την αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φτάσαμε τόσο μακριά, αλλά αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα αριθμιστικό πλαίσιο μοναδικό για την ε, εισδοχή ε, τρίτων, ε, υπηκών τρίτων χωρών ε, που, έχουν, που είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι και πρέπει να πω πως παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως υπάρχει πρόβλημα, εμείς δεν βλέπουμε υπάρχει κάποιο εμπόδιο οικονομικό να υπάρχουν εθνικά συστήματα τα οποία θα συνεπάρχουν με το Ευρωπαϊκό Σύστημα της Γαλάζιας Κάρτας. Η Κομισιόν δεν έχει πιστεί και μίλησε για, μια, για έναν εξευρωπαϊκισμό αυτού του εργαλείου της μεταναστευτικής πολιτικής καλοδεχούμενο. Τρίτον, το κόστος της γαλάζιας κάρτας είναι υπερβολικά και δεν ε, είναι ελκυστική ούτε για τους εργα... εργοδότες, ούτε για τους ενδεχόμενους δικαιούχους, ούτε για τα κράτη-μέλη και τις δικής τους. Και επίσης, επειδή τα κατόφλια στους μισθούς έχουν μειωθεί αρκετά, επίσης, τέταρτον, θεωρούσαμε πως τα ε, εργασιακά δικαιώματα που χορηγεί αυτή η γαλάζια κάρτα ε, δεν, ε, δεν είναι αρκετά πως και αυτό δικαιολογεί το γεγονός πως δεν χρησιμοποιείται πιο ευρέως και για την οικογενειακή επανένωση να σας πω πως ε, αυτό που ε, εξετάσαμε είναι κατά πόσο χρειάζεται αυτό και αν θα πρέπει να είναι πιο εύκολο ολόκληρη η οικογένεια να μετακινείται σε άλλο κρατό μέλο. Γενικά η μεταρρύθμιση είναι καλή, ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Η διαδικασία και να σα πω καταρχήν πω είμαι ε, τμήμα και μέλο τη ομάδα εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να σα πω πω η όλη διαδικασία ήταν αρκετά εξαντλητική. Και βλέπω όντω πω η πρόταση ε, συμπεριλαμβάνει πολλά από τα στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων και που ακούστηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Τρία σημεία κλειδιά είναι σε εκκρεμότητα, είναι προβληματικά. Η γαλάζια κάρτα έχει δοθεί μόνο όταν υπάρχει ε, προσφορά θέσης εργασίας ή ε, σύμβαση και αυτό σημαίνει πως είναι μόνο οι πολυεθνικές που μπορούν να το κάνουν, που πηγαίνουν και ψάχνουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται στο εξωτερικό, που δεν μπορούν να κάνουν μικρομεσές, οι οποίες θα χρησιμοποιούσαν ένα μηχανισμό που θα εξασφάλιζε πως οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε αυτές και όχι πως θα πάνε στη χώρα τους να τους βρουν, δηλαδή ένα είδος αντιστήχησης ε, των διεθνών προσλήψεων που θα είναι πιο απλό θα επανέλθω σε αυτό και επίσης άλλο πρόβλημα είναι πως περιορίζεται στους υψηλά ε, εξειδικευμένους εργαζομένους. Αυτό είναι η γαλάζια κάρτα, αλλά δεν είναι επαρκές. Τρίτον, δεν δίνει ε, πρόσβαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακόμα 28 γαλάζιες κάρτες που έχουν ένα ενιαίο πλαίσιο ρυθμιστικό, αλλά είναι 28 διαφορετικές, 25 θα έλεγα κάρτες, γιατί υπάρχουν τρει χώρες που δεν ε, είναι στο σύστημα. Και το τέταρτο πρόβλημα είναι πως πρόκειται μόνο για πρόταση. Και μένει να δούμε πώς θα υποδεχτούν την πρόταση αυτή το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και αν υπάρχει ο κίνδυνος, όπως έγινε το 2001 με την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα αυτό, πως δεν θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και δεν θα καταλήξει στο ε, το αποτέλεσμα. Εκτός από την γαλάζια κάρτα, κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί, με λεπτομέρειες αν το επιθυμείτε, είναι τρία ζητήματα τα οποία θεωρώ πως είναι ζωτικά. Καταρχήν, σε ποιο μέτρο το θεματολόγιο της Ευρώπης για την μετανάστευση ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχει η Ευρώπη για εργασιακή μετανάστευση. Και όπως είπα πριν, δεν ανταποκρίνεται, αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν λαμβάνει υπόψη την εργασιακή μετανάστευση από τρίτες χώρες ανειδίκευτων εργατών και παρόλα αυτά όταν κοιτάμε τη μελέτη ε, βλέπουμε πως όλες οι μαρτυρίες που έχουμε και τα τεκμήρια που έχουμε για τις ανάγκες σήμερα και στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ότι λείπουν οι εξειδικευμένοι εργάτες, αλλά λείπει ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και να σας δώσω κάποιους αριθμούς. 12 από κάθε 20 σημεία συμφόρησης που βρίσκουμε είναι σημεία συμφόρησης γιατί δεν υπάρχει ακριβώς ανειδίκευτος εργάτης για να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη. Άρα λοιπόν δεν καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς. Δεύτερον, αναλύοντας τις ανάγκες που υπάρχουν και τις μελλοντικές ανάγκες, δημιουργείται η εντύπωση πως πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει η πολιτική εργασιακή μετανάστευση ε, τη στιγμή που θα κληθεί να ανταποκριθεί σε εργασίε ανάγκε που θα έχουμε. Παρόλα τα όσα είπε σήμερα ο κύριο ε, Αβραμόπουλο, επίτροπο, πριν από μια ώρα, αυτή τη στιγμή στι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο μακροπρόθεσμο μοντέλο στο οποίο αναφέρθηκε. Εμείς ε, αναφερόμαστε σε αυτό το μακροπρόθεσμο μοντέλο, αλλά ποια είναι τα στοιχεία που το πλαισιώνουν. Έχουμε κάποια καινούρια στοιχεία. Έχουμε το refit, που είναι η μεταρρύθμιση του πλαισίου και η εξέταση καταλληλότητας αυτού στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής. Υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις ε, ε, πολιτικές που δίνονται για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος της μεταναστευτικής πολιτικής που θα χαράξουμε. Και νομίζω ότι αυτό έχει μία εξήγηση που όλοι γνωρίζετε. Είναι πόσο πολιτικά ευαίσθητο είναι το θέμα το μεταναστευτικό και επίσης υπάρχει και μια νομική και ένας νομικός ε, λόγος και κόλλημα είναι εθνική αρμοδιότητα να ρυθμίσουν την είσοδο των υπηκών τρίτων χωρών. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αυτό το μοντέλο, το νέο μοντέλο της νόμιμης μετανάστευσης που υποσχέθηκε ο πρόεδρος Γιούγκερ εδώ ακριβώς στο κοινοβούλιο ε, τη στιγμή του διορισμού του. Και για την ε, εργασιακή πολιτική και τη μεταναστευτική εργασιακή πολιτική για ανειδίκευτους εργάτες, φαίνεται πως η μεταναστευτική πολιτική θα αντικατασταθεί από την ενσωμάτωση, την πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Εμείς στο δικό μας Policy Center κάνουμε μια μελέτη για το θέμα αυτό και σχεδόν έχουμε τελειώσει, αλλά δεν θα πρέπει εδώ να τον μπερδεύουμε με τη μεταναστευτική πολιτική. Και αυτός είναι ο κίνδυνος σε αυτό το συγκεκριμένο ε, πλαίσιο στην Ευρώπη σήμερα, πού διατρέχουμε. Δεν Μέχρι ποιου σημείο μπορούμε να πούμε πως η βασική σύσταση της μελέτης μας ήταν να πούμε πως η Ευρώπη χρειάζεται μια μεταναστευτική εργασιακή πολιτική η οποία ε, θα είναι ολοκληρωμένη και θα ανταποκρίνει τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Γιατί μετά τις τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζεται αυτή η παράδοξη κατάσταση, ε, η αντίφαση μεταξύ των αναγκών που έχουμε για μετανάστευση εργασιακή λόγω των δημογραφικών τάσεων στην Ευρώπη και από την άλλη έχουμε την έλλειψη εργαλείων που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτή την ενσωμάτωση μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής. Θεσμικά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι είναι η DG Home που για την εργασιακή μετανάστευση είναι αρμόδια και όχι η DG Employment. Ενώ είναι θέμα ε, ώρας εργασίας. Δεν είναι θέμα ε, η ένταση ε, μεταξύ του. Θα πάμε σε μια ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κατάργηση των συνόρων κτλ. Και με την αυξανόμενη ε, ολοκλήρωση αυτών των εργασιακών πολιτικών με τους περιορισμούς που έχουν ή θα διατηρηθούμε με 28 διαφορετικές αγορές εργασίας. Εν πάση περιπτώσει η νέα πρόταση οδηγίας για για την γαλάζια κάρτα δύσκολα θα φέρει αυτά τα ταλέντα που θέλει η Ευρώπη. Γιατί δεν είναι η απόκριση στα διαρθωτικά ερωτήματα που κάνουν την Ευρώπη να μην είναι τόσο ελκυστική όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Αμερική κτλ. Η ΕΠΑ. Είναι διαφθορτικοί λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν κάποιοι με το οικονομικό μοντέλο που έχουμε ή διαφορές μισθών για παράδειγμα για τους ε, που πληρώνουν ε, στους εργαζόμενους ή ο κατακαιρματισμός ο γλωσσικός και βέβαια η έλλειψη ε, του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που νόμιμα διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να κλείσω και να μην καταχραστώ το χρόνο σας, στην τελευταία διαφάνεια έχουμε τις 12 αναλλακτικέ που θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτή η πολιτική, στις οποίες εμβαθύνουμε στη μελέτη μας. Κάποιες έχουν να κάνουν με την διατησία και διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας για τα εργαλεία που έχει ήδη διαθέσιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και για το σχέδιο σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω κάτι να πω. Τους μηχανισμούς εισόδου ή διάβλους εισόδου για τους ε, ξένους ε, ε εργαζομένους, ε, αλλοδαπούς εργάτες κτλ. Και πώς μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το απόθεμα ε, μεταναστών ε, εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σχόλιο πολύ γρήγορο, γιατί έχουμε αυτά τα 12 στοιχεία και θα μπορούσα να τα σχολιάσω αλλά μόνο να τα διαβάσω θα μου πάρει 12 λεπτά, οπότε δεν θα το κάνω. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια, μια ανάγκη να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική στην αγορά εργασίας της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα είναι να συγκολήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα 12 κράτη-μέλη. Και κάτι που ήταν πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι τρεις από όσους πήραν το λόγο για το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις είπαν πως υπάρχει το θέμα της, ε, των στατιστικών στοιχείων, της ενημέρωσης ε, και της γνώσης. Εδώ έχουμε το, ε, την κομμάτι της αλυσίδας που λείπει και εμείς Μαζί με το Ίδρυμα Μπερτέλες μας και με, την, ε, με το δικό μας Policy Center μιλάμε για ανάγκη ε, ενσωμάτωσης των προσφάτων προσφύγων και των ετούντων άσυλο στην αγορά εργασίας. Κάναμε μια γρήγορη μελέτη σε νέα κράτη-μέλη και αυτό που κάναμε ήταν κυρίως προσπαθήσαμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες για το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί και τι γίνεται. Μια γρήγορη απογραφή δηλαδή των μέτρων στήριξης που έχουν ε, ισχύσει στα εννέα κράτη που εξετάσαμε. Το βασικό συμπέρασμα και η μελέτη αυτή θα είναι έτοιμη και θα δημοσιευτεί σε δύο εβδομάδες είναι πως δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γνωρίζουμε ελάχιστα για το προφίλ, για παράδειγμα, ή για τη διάστρωση αυτών των ομάδων, όπως είπε η Ευρωβουλευτής, για τις ομάδες που καταφθάνουν κυρίως τους ε, πρόσφυγες και όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο παιδείας, δεν ξέρουμε τι, ποια είναι η επαγγελματική του σταδιοδρομία, δεν ξέρουμε τίποτα. Και έχουμε απλώς κάποια ε, μερικά ε, στοιχεία, αλλά δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Και αυτό επηρεάζει τα μέτρα που εφαρμόζουμε. Και στα πλαίσια του σχέδιου δράσης για την ενσωμάτωση ε, νομίζω ότι έχει φτάσει πια η στιγμή να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε μια καλύτερη δημιουργία ε, πληροφοριών ε, και μια καλύτερη ενημέρωση γιατί ξέρω πως η Κομισιόν θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο το κόστος για να το καταφέρουμε. Τόσα κονδύλια χρησιμοποιούνται για άλλα πράγματα. Και ίσω το νέο αυτό δίκτυο στην Ευρώπη για την ενσωμάτωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έμβριο που θα γεννήσει περισσότερες προφορίες, περισσότερη έρευνα, περισσότερα στοιχεία. Και μια τελευταία παρατήρηση σημαντική για κάποιο άλλο από τα μέτρα. Δύο από τι εναλλακτικέ λύσει που αναλύονται είναι και το μοντέλο της ε, πρόσκλησης με ε, προσυνέντευξη των όσων θα φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εκεί εξηγούμε γιατί δεν θεωρούμε πως το σύστημα αυτό, το οποίο ε, στον Καναδά λειτουργήσε κάπως καλά, δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα σε άλλα γιατί τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εργασία και Μετανάστευση έχουν ε, κοινωνικά κράτη και το γεγονός πως έχεις αυτό το ε, σύστημα πόντων και το κράτος πρόνοιας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και πιστεύουμε πως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα που θα έχει να κάνει περισσότερο με την προσφορά που θα επιτρέπει στους υποψηφίους να ψάξουν να βρουν δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, μέσω μιας θεώρησης ε, βραχυπρόθεσμης που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ψάξουν δουλειά για άνθρωπους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ και που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Σταματώ εδώ. Και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάρτιν. Κυρία Ζίπελ, πρώτη. Very much. I would like to ask several questions. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να, ρωτήσω, να διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πως τονίσατε πως η με την παράνομη μετανάστευση σε θέσεις εργασίας θα χρειαζόμαστε μόνο ψηλά καταρτισμένους ανθρώπους, αλλά μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα παρουσιάζεται επίσης η ανάγκη εργαζομένων με διαφορετικά επίπεδα προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ πλήρω πως αυτό ισχύει. Ταυτόχρονα, για να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός και κυρίως ο αθέμητος ανταγωνισμός με τους πολίτες, πρέπει να διασφαλιστεί πως οποιοδήποτε νεο, νεοαφιχθής στις εργασίες μας έχει δίκες συνθήκες εργασίας. Αυτή είναι η προϋπόθεση βέβαια. Για να συγκρίνουμε την κατάστασή μας με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύω πως αυτό δεν είναι ακριβώς δίκαιο, επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον προσπαθούμε να έχουμε ένα καλό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο έχει κάποιες αντίψεις σε σχέση με ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κάποιες ελλείψεις σε σχέση με αυτό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν συμφωνώ πως οποιαδήποτε παράνομη μετανάστευση προς την αγορά εργασία. θα πρέπει να προσφέρεται για όλα τα επίπεδα προσόντων. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο σε πρώτο βαθμό μπορούμε να συμφωνήσουμε να επιτρέψουμε την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας επειδή οι συνθήκες στα κράτη-μέλη είναι πολύ δύσκολες. Καθώς είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς εργοδότες, αλλά επίσης ως προς κάποιες άλλες συνθήκες πλαισίου. Γι' αυτό και πιστεύω πως είναι απαραίτητο να πούμε πως φυσικά πρώτα πρέπει να δούμε την κατάσταση των δικών μας πολίτων και τον βαθμό στον οποίο χρειάζεται κατάρτιση εκεί. Πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τους ετούντες άσυλο που βρίσκονται στις χώρες μας, τι προσόντα έχουν, τι μπορεί να γίνει για την καλύτερη ένταξή τους στους χώρους εργασίας μας και τότε μπορούμε να ελέγξουμε ποια πρόσθετα προσόντα χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι κάτι πολύ, αυτό διαφέρει πάρα πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, από περιοχή σε περιοχή. Και αυτό και η ερώτησή μου είναι, μπορείτε να συμφωνήσετε πως χρειάζεται να, πάρουμε ένα διάμεσο, να κάνουμε ένα διάμεσο βήμα, έτσι ώστε οι μετανάστες και οι εργαζόμενοι να μην έχουν σε ανταγωνισμό σε ορισμένα μέρη, επειδή αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, επειδή αν χρειάζεται να έχει κανείς μια σύμβαση εργασία, τότε αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκ μέρους μεγάλων επιχειρήσεων. Αλλά αυτό δεν ισχύει πλήρω. επειδή πιστεύω πως κάποια κράτη-μέλη που ψάχνουν ήδη πρόσθετου εργαζόμενους αναλαμβάνουν τα ίδια δράση. Η Γερμανία το κάνει, ψάχνει σε άλλα κράτη για εργαζόμενους και προσπαθεί να βρει στις τρίτες χώρες κατά πόσο μπορεί να βρει πρόσθετους εργαζόμενους εκεί. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση για οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν και στις τρίτες χώρες και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καταστούν προσβάσιμες και στις τρίτες χώρες. Είναι ζητήματα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αποτελεί τμήμα της μελέτης σας να βρούμε κατά πόσον χρειάζονται κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα ή κατά πόσον αυτό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών λόγω των δυνατοτήτων που έχουν αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσω στη συζήτηση, επιτρέψτε μου να, να καλωσορίσω κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης που εισήλθαν στην αίθουσα πριν. Είστε καλοδεχούμενοι στη συζήτηση. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Πινέλη. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα επαναλάβω ε, μια ερώτηση που έκανα και προηγουμένως προς την Επιτροπή, αλλά δεν έλαβα για αυτήν καμία απάντηση. Μπορεί ίσως να μου απαντήσετε εσείς. Αφορά τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης, ένταξης, πρόνοιας και εργατικού δικαίου. Ο λόγος που σας απευθύνομαι είναι γιατί μιλήσατε για τις ανάγκες για εργασίες υψηλών προσόντων από τις μεγάλες εταιρείες σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες. Δεδομένων των στοιχείων που μας δώσατε. Πώς μπορούμε να δούμε αυτόν τον ανταγωνισμό ε, υποβάθμισης το χώρο εργασίας των κρατών μελών. Πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε τον φόβο που έχει διαδοθεί σε διάφορα κράτη-μέλη. Φόβο για αυτήν την ε, τάση υποβάθμισης. Την ε, πιθανότητα να χάσει κανείς δικαιώματα. Δικαιώματα της Ευρώπης στην πρόνοια. Να θυμίσω ότι το εργατικό δίκαιο στα κράτη-μέλη καθορίζεται στην ουσία σε επίπεδο ευρωπαϊκού εξαμήνου και όλοι οι νέοι κανόνες έχουν πλέον μια σαφή τάση προς τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας με την ολοένα και μεγαλύτερη διεύρυνση δικαιώματος απολύσεων, απελευθέρωσης των απολύσεων. Θα ήθελα τουλάχιστον εσεί να μου δώσετε μια απάντηση και κλείνοντα να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφο Ζήπελ. Για, το, για τη δυσκολία να συγκρίνουμε διαφορετικές πραγματικότητες των κρατών μελών στην Ευρώπη είχαμε επίπεδα κοινωνικής προστασίας μάλλον υψηλά τα οποία όλο και λιγότερο ισχύουν βέβαια χωρίς πρόβλημα αλλά θα το σχολιάσετε κι εσείς ελπίζω. Ευχαριστούμε κυρία Λάουριστην. Ευχαριστώ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πραγματικά την απίλαυσα. Και για τα όσα κάνει το κέντρο σας. Για τα θέματα ένταξης στην Εστονία. Είναι θέματα που μας να απασχολήσει από πολύ καιρό και στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία μας πώς θα εντάξουμε αλόγλωσσους και αλλοδαπούς στη χώρα μας. Η ένταξη πικών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας εδώ και καιρό έχουν, έχει δημιουργήσει πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά στο κέντρο σας, σας έχουν φανεί χρήσιμα. Και μιλάμε στην φάση μιας μεγάλης κρίσης προσφύγων. Οι άνθρωποι που έρχονται από τρίτες χώρες ε, πολλές πρέπει να προσαρμοστούν σε μια τελείως νέα κατάσταση. Όλη η δουλειά που έχει γίνει εκ των προτέρων ε, και με ανθρώπους που είναι ήδη ενταγμένοι ή ανθρώπους που μεταναστεύουν ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ένα κατός μέλος σε άλλο κατός μέλος. Φαίνεται σαν να ζουν σε παράλληλους κόσμους, σαν να είναι διαφορετικές πραγματικότητες. Το ερώτημα είναι πού μπορούν να συγκλίνουν όλα αυτά. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι η αγορά εργασία είναι μία. Και ότι αυτές οι διαφορετικές ροές, παλιές νέες, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά. Ποια είναι η δική σας θεώρηση, βλέποντας το εργατικό δίκαιο και όλα αυτά τα ζητήματα. Αν δούμε αυτό τι μπορεί να γίνει σε μία πενταετία. Τι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ανταγωνισμό, το εργατικό δίκαιο, το κόστος της εργασίας, τους κανονισμούς, τους κανόνες μάλλον για την απασχόληση. Μας κοστίζει πάρα πολύ αυτή η κατακαιρματισμένη προσέγγιση, αυτή η διάσπαση. Η επιθυμία να συγκλίνουν οι απόψεις μας και οι ματιές μας, αλλά και η διάθεση προστατευτισμού στην αγορά εργασίας είναι ακόμη πολύ ισχυρή. Ε, κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι όλο μιλάμε για ανοιχτή κοινή αγορά εργασία στην Ευρώπη και ότι αυτό δεν ισχύει καθόλου. Δείτε τι γίνεται στην Γαλλία και το καθεξής. Ποια είναι η δική σας θεώρηση. Τι στάση πρέπει να τηρήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα, έχοντα υπόψη θα συμβεί στην αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πέντε χρόνια. Κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη μελέτη και ευχαριστούμε και για την ειλικρίνειά σας, την ευθυκρισία σας. Τα λέτε πραγματικά όπως είναι τα πράγματα, κοφτά. για κάποια από τα σχόλια που κάνατε για τις ελλείψεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πόσο η ευελιξία αφήνεται στα κράτη-μέλη για να αποφασίσουν. Όντω, η γαλάζια κάρτα ήταν ένα από τα ωραιότερα εγχειρήματα και παραδείγματα, αλλά το πρόβλημα που δημιουργεί η απουσία ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη να έχουμε καλύτερα στατιστικά δεδομένα ε, και ποιοτικά, όλος ιδιαίτερος ποιοτικά για αυτές τις δύο πτυχές, είναι σημαντικό. Είναι μέρος των φόβων και των προκαταλήψεων που υπάρχουν. Η απουσία τέτοιων πολιτικών οδηγεί σε μείωση των ένομων οδών ε, για τη μετανάστευση των εργαζομένων συμφωνείτε με αυτήν την άποψη στην μελέτη σας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα περισσότερα για το θέμα της σύγχυσης. Σύγχυσης μεταξύ μετανάστευσης εργαζομένων και προσφύγων. Ε, εάν μπορούσατε να το σχολιάσετε λίγο παραπάνω. και σημείωσα μεταξύ των προτάσεών σας την στοχευμένη νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών. Το βρίσκω σημαντικό μεταξύ άλλων διότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε την έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ πραγματικότητας ε, της πολιτικής της Ευρώπης και των αναγκών που υπάρχουν. Νομίζω όλοι διαπιστώνουμε, αλλά εγώ όλος ιδιαίτερος στη Γαλλία, ότι πολύ μεγάλο μέρος της μετανάστευσης γίνεται μέσω της επανένωσης των οικογενειών, διότι η κανονική μετανάστευση έχει σχεδόν σταματήσει, έχει κλείσει η βρυσούλα και έχει στερέψει η πηγή, οπότε υπάρχουν ε, μετανάστες εργαζόμενοι σε ε, μη ε, με χαμηλό προσόντων επαγγέλματα, με όσα έχουν να κάνουν με την εστίαση, τις υπηρεσίες προς τον συμπολίτη, Θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε αν μπορείτε. Έχουμε μεγάλη τέτοια ζωή και για την αναγνώριση των πτυχίων. Την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων. Μου φαίνεται πολύ σημαντικό διότι μιλήσαμε για χαμηλών προσόντων επαγγέλματα, αλλά βρίσκουν μετανάστε υψηλότατων προσόντων που δεν έχουν επιλογή. Παρά να πιάσουν μια τέτοια δουλειά, γιατί είναι η μόνη που του προσφέρεται. Εάν μπορείτε λοιπόν να το αναπτύξετε λίγο, θα με ενδιαφέρετε. Κυρία Βεργιά, ευχαριστούμε. Και τώρα να σας δώσω πάλι το λόγο, κύριε Μάρτιν, για τις απαντήσεις σας. I will respond in English that I understand is the more or less the common, the most common language uh, of the uh, uh, members of the Parliament who have made questions. Well, first thing. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Πρώτον, όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ της πολιτικής της αγοράς εργασίας και της πολιτικής για τους πρόσφυγες. Η πολιτική για την αγορά εργασίας απευθύνεται στην αγορά εργασίας. Έχει ένα οικονομικό υπόβαθρο και δεν ασχολείται παραδείγματος με ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δικαιο ένταξης των προσφύγων βασίζεται σε διεθνείς δεσμεύσεις και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και το να μίξει κανείς τα δύο αυτά θα δημιουργήσει πολλές στρεβλώσεις και πιστεύω από πολλές απόψεις. Παραδείγματος χάρη θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο απόδειγμα. Όλοι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι, μέχρι και η Επιτροπή, με την προοπτική του να ανοίξει η μπλε κάρτα για αυτούς που δικαιούνται διεθνή προστασία και έχουν τα προσόντα. Πολύ ωραίο αυτό, αλλά σκέφτηκε ποτέ κανεί τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Αυτό σημαίνει κατά βάση πως χώρες όπως η Πολωνία, η Εσθονία ή η Ελλάδα ή ελλαδα η ισπανια που δεν έχουν πολύ δυναμικές, που δεν έχουν πολύ δυναμικές αγορές για εργαζόμενους με υψηλά προσόντα, θα ανοίξουν για λίγους υψηλά καταρτισμένους πρόσφυγες, παραδείγματος χάρη, επειδή θα, κατα... θα, κατα θα καταθέσουν την αίτηση για μια μπλε κάρτα στη Γερμανία και η Γερμανία θα χαρεί πάρα πολύ να πάρει τους ε, πρόσφυγες αυτές οι οποίοι έτσι γίνονται οικονομικοί μετανάστες. Η προσέγγιση φαίνεται ορθολογική, αλλά ενέχει τον κίνδυνο στρεβλώσεων δεύτερων ισχύση μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ευρώπης. Πιστεύω πως παρανοήθηκα. Συμφωνώ απόλυτα πως δεν μπορούν να συγκριθούν και αυτή είναι η κύρια ανησυχία μου όταν ακούω την Κομισιόν η κύρια ιδέα για την πολιτική, για την νόμιμη μετανάστευση είναι η θέσπιση της εκδήλωσης συμφερόντων κοντά στο καναδέζικο μοντέλο. Στον Καναδά όμως το ποσοστό των νόμιμων μεταναστών στην αγορά εργασίας είναι υψηλότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως τα κράτη πρόνοιας, ιδίω για αλλοδαπούς, δεν είναι τόσο εξελιγμένα όσο στην Ευρώπη και οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη λύση από το να εργαστούν. Πολλοί από αυτούς, εάν βρίσκονταν στην Ευρώπη, δεν θα εργαζόταν. Δεν θα εργάζονταν επειδή θα μπορούσαν να επωφεληθούν, δόξα τω Θεώ πρέπει να πω, από το τις παροχές του κράτους πρόνοιας. Γι' αυτό και αυτό που θέλω να πω κυρίως είναι πως πρέπει να προσέχει κανείς πάρα πολύ κατά τη σύγκριση διαφόρων κοινωνικών και νομικών συστημάτων κατά την χρήση των ίδιων εργαλείων. Στην Ευρώπη έχουμε πολλούς υψηλά καταρτισμένους ανέργους. Εγώ είμαι από μια χώρα με πολύ υψηλή ανεργία αποφύτων εξειδικευμένων αποφύτων πανεπιστημίου έως 50% στους νέους, 30% στους απόφυτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι άνεργοι. Με ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να φέρουμε στην ευρωπαϊκή αγορά εργασία, παραδείγματο χάρη, την ίσιου απόφυτους οι οποίοι επίση μπορεί να γίνουν άνεργοι απόφοιτοι, όπως είναι ήδη η συνομιλική του στην Ισπανία. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την παροχή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε υπηκόους των χωρών. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έτσι κι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επειδή τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα για, την, για τον προσδιορισμό των τον αριθμό στους οποίους παρέχεται η πρόσβαση αυτή. Σίγουρα θα είναι μια σταδιακή προσέγγιση, δεν υπάρχει άλλη νομική δυνατότητα. Κατόπιν αυτό θα θέλω να πω επίσης πως όπως τα κρατημένη μελη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχθηκαν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας όλων των υπηκών των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να γνωρίζουν τα επαγγελματικά τους περιγράμματα ή τις ηθαγένειές τους. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει επίσης για την ελεύθερη κυκλοφορία επικών τρίτων χώρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει οικονομικό νόημα. Θα αναφερθώ σε μια ερώτηση που θέσατε, κάποιο από τα μέλη του Κοινοβουλίου την έθεσε, το ζήτημα της αναγνώρισης προσόντων. Πιστεύω πως και πάλι η αναγνώριση προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται κατά βάση στην ευρωπαϊκή Ιθαγένεια σε αυτή την ιδέα και όχι σε οικονομικούς λόγους. Και αυτό οδηγεί σε αντιφάσεις, πως δηλαδή υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους σε ένα κράτος μέλος, αλλά μετά δεν αναγνωρίζονται στο άλλο. Και είναι απίστευτο αυτό. Εγώ ως Ισπανός, εάν κάνω το διδακτορικό μου στο London School of Economics, τότε υποχρεωτικά αναγνωρίζεται στα άλλα κράτη-μέλη. Όχι αυτόματα, αλλά έχω το δικαίωμα να αναγνωρίσω εύκολα αλλά ένας υπήκος ενός τρίτου, μιας τρίτης χώρας με το ίδιο πτυχίο, το ίδιο διδακτορικό στο London School of Economics δεν έχει το δικαίωμα αυτό το, της αναγνώρισης του διδακτορικού του. Αυτό από οικονομικής άποψης δεν έχει το παραμικρό νόημα. Εμποδίζει υψηλά καταρτισμένους υπηκόστριτων χωρών να έρθουν στην Ευρώπη. Οπότε είτε έρχονται επειδή είναι όντω πάρα πολύ υψηλά καταρτισμένοι, οπότε βρίσκουν μια καλή λύση, μια καλή προσφορά, ή δεν έχουν άλλη εναλλακτική. Όσον αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Σηκώνω πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Αλλά καθώ εργάστηκα πολύ επί του πεδίου για την πολιτική αγορά εργασία. γνωρίζω πώ είναι η αγορά εργασία. Είναι πολύ επί οτιδήποτε δεν φέρνει νέους εργαζόμενους στους εργοδότες δημιουργεί μειονεκτήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά και στις προτάσεις της Επιτροπής δεν είδα καμία την παραμικρή προσπάθεια αντιστοίχησης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Υπήρξε η ιδέα διεύρυνσης του ευρωσυστήματος σε τρίτης χώρες. Δεν το άκουσα ποτέ, ίσως και επιλεκτικά. Όποτε τι θέλετε, το ζήτημα αυτό, τα κράτη-μέλη λένε όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Και αυτό αποτελεί επίσης ένδειξη για το ότι δεν ε, αναπτύσσουμε μια πολιτική περιεργασιακής μετανάστευσης αλλά ότι κάνουμε μεταναστευτική πολιτική ανεξάρτητα από την πολιτική για την εργασία. Όπου μπαίνουν στο παιχνίδι βραχυπρόθεσμε πολιτικές σκέψεις, οι οποίες είναι νομιμοποιημένε, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη οικονομικά ορθολογικέ. Όσον αφορά το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ μετανάστευσης, ένταξη και, ένταξης και Γι' αυτό θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ένα-δύο Είναι ένα πολύ περιπλοκό ζήτημα, αλλά θα είμαι σαφής και θα το σύνδεσω με την προηγούμενη ερώτηση. Πιστεύω πως ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε ή τουλάχιστον για να αναχαιτήσουμε ή για να καταπολεμήσουμε την κατάκριση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας είναι περισσότερη, η περισσότερη ένταξη των αγορών. Αλλιώς χάσαμε ήδη ένα μεγάλο ζήτημα. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε καν μία αγορά εργασία στην Ευρώπη. Και θα βάλει πολύ καιρό μέχρι να εξελιχθεί αυτή. Όσον αφορά την κοινή τιμή, συμφωνήσαμε να θεσπίσουμε το ευρώ πριν την εναρμόνιση των συνθήκων εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη και τώρα θα χρειαζόταν μια οικονομική επανάσταση για να το κάνουμε. Οπότε η Ευρώπη με αυτούς τους όρους δεν θα γνωρίσει ποτέ μια εντελώς ενιαία αγορά εργασίας. Αλλά όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και την ελεύθερη κυκλοφορία, όχι μόνο για τους υπηκόους των κρατών μελών, αλλά και για τις τρίτες χώρες που ζουν μόνιμα στα κράτη-μέλη, πιστεύω πως είναι μια ξεκαθαρή τάση και μια ξεκαθαρή ανάγκη, όχι μόνο όσον αφορά την εργασιακή μετανάστευση, αλλά γενικότερα με όρους προστασίας του κεκτημένου του κράτους πρόνοιας. Είμαι πολύ, σαφό, σα, πολύ σαφής προς αυτό. Δεν θα μπω περισσότερο εις βάθος για λόγους χρόνου. Όσον αφορά την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, Έχουμε ενδείξεις από την έρευνα από εννέα χώρες, επίσης πρακτικές ενδείξεις, η Σουηδία, η Γαλλία, η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, η Εστονία δεν ήταν, και το Ηνωμένο Βασίλειο, συγγνώμη το ξέχασα. Το συμπέρασμά μας είναι πως η ένταξη προσπήγων και τούτων άσελος στην αγορά εργασίας είναι ένα πολύ περίπλοκο και πολύ δύσκολο ζήτημα δεν είναι ένα μηχανικό ζήτημα ε, αναγνώρισης δεξιοτήτων. Υπάρχει το ζήτημα των κινήτρων. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Καμία χώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, σίγουρα όχι η Σουηδία πάντως, δεν τα κατάφερε να βρει την, ε, να βρει τον κατάλληλο τρόπο για αυτήν την ένταξη αν κοιτάξει κανεί την αγορά εργασία τη Σουηδία, θα δει πως υπάρχουν πως έχουμε επιστροφές σε προηγούμενα μοντέλα. Έχουμε υποχρεωτικά εθελοντικά προγράμματα, δημοτικά προ προγράμματα, κανένα από αυτά δεν λειτουργήσε απόλυτα. Φυσικά οι πρόσφυγε εντάσσονται στην αγορά εργασία, αλλά εντάσσονται αργότερα από τους μετανάστες και ακόμα αργότερα από τους ντόπιου. Είναι προφανές αυτό και είναι αποδεδειγμένο. Και αυτό μάλλον θα συνεχίσει ως έχει. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια πολιτική ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασία, αλλά επίση μια πιο φιλόδοξη πολιτική η οποία θα αποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας το οποίο δεν μπορεί να γίνει δια της πολιτικής ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Όπως και να έχει, για να απαντήσω την ερώτηση, Πολύ προσοχή έχει δοθεί σε αυτά που κάνουν επί χρόνια η Σουδία, η Δανία. Αυτό που έκανε τα τελευταία χρόνια επίσης η Γερμανία. Αλλά δεν βλέπω, θα έλεγα, δεν βλέπω ότι διαδίδονται διδάγματα, ίσως επειδή δεν έχουμε συστηματική ανάλυση των αποτελεσμάτων της εργασίας και της έλλειψης και, και της αδυναμίας των εθνικών και υπερεθνικών παικτών να συλλέξουν δεδομένα για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες ωστόσο λειτουργούν κυρίως αθόρμητα. το, το ζήτημα της νομιμοποίησης, θα είμαι σαφής, ένα οικονομικό πρόταγμα πίσω από αυτή την επιλογή είναι πολύ απλό. Εάν οι παράτυποι μετανάστευς έχουν μία δουλειά, δεν θα κοστίζουν. Τότε πρέπει να ληφθούν δύο μέτρα. Το πρώτο είναι η αποστολή των επιθεωρητών εργασίας για την για να ελέγχεται τη τήρηση των ελάχιστων προτύπων εργασία και το δεύτερο είναι η νομιμοποίησή τους. Κατά βάση νομιμοποιούμε έναν, μηχανισμό ο οποίος δημιουργεί και διατηρεί την επισφάλεια και για αυτόν τον άδικο ανταγωνισμό με μη χαμηλά καταρτισμένους ντόπιου εργαζόμενους. Αυτή είναι η λογική πίσω από αυτό και λειτουργήσε καλά και μάλιστα στη χώρα μου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμάμαι το 2005 η Ισπανία δέχτηκε πολύ κριτική και χαίρομαι που επιτέλους μπορώ να πω κάτι καλό για την μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Η Ισπανία έλαβε πολύ κριτική για την νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών. Και ενώ σήμερα θεωρείται επιτυχία. Έχουν ενταχθεί. Μα και βέβαια. Αλλά όταν ήρθε η κρίση προέκυψαν υψηλή υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά αυτό αποτελεί μέρος της αγοράς εργασίας. Μετά την ομοποίηση αυτή και την κρίση στην αγορά εργασίας, δεν βλέπω υψηλότερε πολιτικέ ή χειρονικέ εντάσει γύρω από το ζήτημα τη μετανάστευση από ό,τι σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. θα, φτάσω, θα τελειώσω εδώ, εάν συμφωνείτε, εκτός αν θέλετε να πω κάτι άλλο. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας, για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και για όλη σας τη δουλειά. Εξαντλήθηκαν τα σημεία τη ημερήσια διάταξη για σήμερα, οπότε κυρίζω τη λήξη τη σημερινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στι 9. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι, για τη συνεργασία σα και για το ενδιαφέρον σα.